γυναίκες και να έχουμε μια καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών δεν είναι μόνο προς όφελος των γυναικών αλλά και για τα δύο φύλλα. Και θα πρέπει και τα δύο φύλλα να φροντίσουν να έχουμε καλύτερη και πιο δημοκρατική νομιμοποίηση στα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τις εκλογές. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συμβάλλει στις εκλογικές εκστρατείες με μια σειρά μέτρων και εκεί θα ζητήσουμε από εσά ως δημοσιογράφοι να παρουσιάσετε, να καλύψετε αυτές τις διάφορες ε, ιστορίες ε, που ε, παρουσιάζονται γιατί ίσως δεν ενδιαφέρονται πολύ για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρονται και οι γυναίκες και οι άνδρες και αυτά θα πρέπει να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I like to... Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιος από εσάς να κάνει κάποια σχόλια, να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στις δύο μιλήτριες. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, να υποβάλω μια ερώτηση προς την Επίτροπο Βάλστρομ. Δίνουμε την εντύπωση ότι, δίνετε την εντύπωση ότι αν οι γυναίκες είναι στη διαδικασία λήψης αποφάσεις, σημαίνει αυτόματα ότι εκπροσωπούνται οι γυναίκες και τα συμφέροντα των γυναικών. Εμείς μπορούμε να φανταστούμε όλες τις χώρες μας πολλά παραδείγματα υψηλά ισταμένων γυναικών πολιτικών που δεν λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα τα θέματα των γυναικών, ε, που δεν είναι. Δεν είναι αυτό μετά, δηλαδή η γυναίκα προσωπεί τα θέματα της γυναικών. Όχι, δεν έχουμε πολλά ε, παραδείγματα. Υπάρχουν ορισμένα καλά προ, παραδείγματα, ίσως σκεφτόσαστε στην ε, ε, χώρα σας, όπου αυτό χρησιμοποιείται σαν ένα ε, παράδειγμα από τη χώρα της ότι οι γυναίκες μπορούν να πάρουν ρατσιστικές αποφάσεις ή κάποιες αποφάσεις που είναι εις των γυναικών. Ναι, αλλά ξέρουμε όμως ότι αν καλύτερα δημοκρατικά εκπροσωπηθούν οι γυναίκες και τα συμφέροντα των γυναικών θα τεθούν επιτάπητος. Αυτό τι σημαίνει ότι αυτά που παραδοσιακά είναι οι εμπειρίες των γυναικών θα προωθηθούν, θα τεθούν στην ημερησία διάταξη. Το ξέρουμε από μια σειρά ερευνών των Ηνωμένων Εθνών και τις στατιστικές των Ηνωμένων Εθνών. Θα μπορούμε έτσι να έχουμε συμπληρωματικές προοπτικές διαδικασία λήψης απόφασης. Δεν είναι ότι αξιολογούμε ότι οι γυναίκες κάνουν πράγματα που είναι καλύτερα ή όχι καλύτερα, αλλά είναι η δική τους εμπειρία, οι δικές τους ιδέες. Μπορούμε να πούμε ότι το 70% του πληθυσμού να μην έχει ψήφο. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλύτερες ιδέες, είναι διαφορετικές γιατί έχουμε τις δικές τους εμπειρίες, τις δικές τους ιδέες, τις δικές τους γνώσεις. Αυτό είναι, αυτό είναι το σημείο κίνησης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε τώρα το λόγο για να υποβάλει κάποια ερώτηση ή να κάνει κάποια παρατήρηση. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι πρωτού. Θέλω να συμπληρώσω κάτι πρωτού σας αφήσω, διότι είμαι εδώ μόνο για το opening, ε, να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω, το οποίο έχει να κάνει με τη συμμετοχή των γυναικών ακριβώς στις ευρωεκλογές και το τι περιμένουμε από τη γυναικεία συμμετοχή. Δεν πρέπει να παγιδευτούμε στην αναζήτηση και στον θαυμασμό μόνο των γυναικών που βρίσκονται στην κορυφή. Διότι αυτό συμβαίνει στη ζωή, συμβαίνει σε όλες τις χώρες, συμβαίνει στα ευρωπαϊκά όργανα, μπορεί να συμβεί ακόμη περισσότερο αύριο, να βρεθούν γυναίκες στην κορυφή. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, το οποίο σημαίνει πολλές θυσίες για μια γυναίκα, που εμείς οι γυναίκες το καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο. Πρέπει να σταθούμε με προσοχή ότι η αλλαγή της κοινωνίας, η αλλαγή των, του τρόπου εργασίας, ε, των πολιτικών οργάνων. Έχει ανάγκη από πολλές γυναίκες σε πολλά επίπεδα. Δεν θα αλλάξουν αυτόματα τα πράγματα αν βρεθούν κάποιες γυναίκες σε μια υψηλή κορυφή. Για μένα κορυφή είναι κάθε επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται αποφάσεις και κάθε επίπεδο έχει ανάγκη από μια κριτική μάζα, όπως τη λέμε, που είναι ένας απαραίτητος αριθμός, οι στατιστικές λένε γύρω στο 30% τουλάχιστον, για να υπάρχει μια πραγματική συμβολή, γυναικεία συμβολή στην παραγωγή αποφάσεων και στην εφαρμογή πολιτικών. Γι' αυτό έχει σημασία αυτό το μήνυμα στι ευρωεκλογέ, γιατί οι ευρωεκλογέ πρέπει να αναδείξουν, όπω μα λέει η έρευνα που θα αναλύσετε στη συνέχεια, ζητούν οι πολίτε 50% των γυναικών. Λοιπόν, με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που 50% θα είναι γυναίκες ε, ευρωβουλευτές, εκεί μπορούμε να περιμένουμε σημαντικά πράγματα. Μακάρι να βρεθούν γυναίκες και στην κορυφή των ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά σημαντικό είναι να βρεθούν πολλές γυναίκες στις επιτροπές, κοινοβουλευτικές επιτροπές, στις αποστολές, σε όλες τις πολιτικές, σε όλες τις εκφράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Ευχαριστώ. Thanks Σας ευχαριστώ πολύ. Μήπως κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Ε, το χέρι σας σας παρακαλώ να σηκώνετε. Παρακαλώ. Η κυρία ροζ Πουλόβερ. Κυρία Επίτροπε, ε, μια ερώτηση προς την κυρία Βάλστρομ θα ήθελα να θέσω. Αναφέρατε το, την Guardian. Εγώ αναφέρομαι σε μια έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εχθές για τις γυναίκες στην πολιτική και διάβασα ότι από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1958 το 58, συγγνώμη, είχαμε 128 γυναίκες που είχαν λάβει θέση ε, συγγνώμη, 128 άτομα που είχαν λάβει θέση ως Ευρωπαίοι Επίτροποι και μόνο 19 γυναίκες. Ο πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν γυναίκα όμως. Μήπως ήγη και να έχουμε και μία γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν ναι, εσείς θα είστε υποψήφια. Ευχαριστώ. Ντανιέλα Μίτσνερ από το Euroactive. Έχετε δίκιο. Από τους Από τους 15 Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο μία ήταν γυναίκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Είναι πολύ ε, περίεργο το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να έχουμε περισσότερες γυναίκες σε υψηλά αξιώματα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν θα είμαι εγώ υποψήφια. Είμαι ήδη 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Θα συνεχίσω με την πολιτική μου πορεία και θα ασχολούμαι με θέματα ισότητας των φύλων με τον ένα με τον άλλο τρόπο, αλλά δεν θα είμαι υποψήφια. Θα μπορούσα όμως κάλλιστα να σας αναφέρω κάποια ονόματα για να σας δείξω ότι υπάρχουν γυναίκες με προσόντα που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιες ε, για τις ε, προεξάρχουσες θέσεις. Αυτό ακριβώς που είπατε είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτή την εκστρατεία η οποία ονομάζεται Δημοκρατία 50-50 και αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές ως υποψήφιες. Ε, θα ήθελα λοιπόν να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λοιπόν κάποια στοιχεία για το ποιος θα θέλατε στην Προεδρία. Δεν έχω έναν αριθμό υποψηφίων που θα μπορούσα να πω ότι μίλησα μαζί τους και θα μπορούσαν να είναι υποψήφιες, αλλά θα μπορούσα κάλλιστα να σας αναφέρω μια σειρά από γυναίκες που είναι ήδη ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Μπαίνοντα, ε, είδα την Ούρσολα Πλάσνικ, την Άννα Διαμαντοπούλα, την ε, Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, η οποία είναι μια έξοχη γυναίκα πολιτικός, την Τάρια Χάλουνεν, ε, την Άγγελα Μέρκελ. Έχουμε αρκετές γυναίκες οι οποίες είναι είτε υπουργοί εξωτερικών ή υπουργοί εν γέννη που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι υποψήφιες και για υψηλότερα αξιώματα. Αλλά είναι αόρατες. Όταν ξεκινάμε τη συζήτηση ξεκινάμε πάντα με τα ε, βασικά ονόματα. Και αυτή ήταν και η επικεφαλίδα του τίτλου που είδα ήταν τρει άντρε για την Ευρώπη. Γιατί τρει άντρε για την Ευρώπη. Οι, μισές γυναίκες, η μισός πληθυσμός Ευρώπης είναι γυναίκε. Γιατί να μην έχουμε λοιπόν και δύο γυναίκε στον ίδιο τίτλο. Δεν είναι μόνο θέμα οι γυναίκες να παρουσιάσουν ονόματα, αλλά και οι άντρες και οι γυναίκες να παρουσιάζονται. Πρέπει να έχουμε ίση εκπροσώπηση και αυτό θα βοηθήσει και τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτό άλλωστε είναι και το σημείο κίνησής να αποχαιρετήσουμε την κυρία Κράτσα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Η κυρία Χάνιμπολ που είναι ε, Βρετανίδα Ευρωβουλευτής από το Εργατικό Κόμμα θα ήθελε να μας πει κάποια πράγματα. Συγγνώμη Μάργαρετ, δεν άκουσα όλη σου την ομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας και όλων όσων κάνεις. Εκείνο που ήθελα να θίξω είναι το εξής. Όσον αφορά στους ευρωβουλευτές, τα πολιτικά κόμματα είναι αυτά που αποφασίζουν και από την πείρα μου στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν γίνεται τυχαία αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν δομές, ε, δεν ξέρω, μπορείτε να τις αποκαλέσετε πώς θέλετε. Νομίζω ότι και στη Σουηδία ένας από τους λόγους που είσαστε εσείς τόσο επιτυχημένοι είναι γιατί κάνετε κάτι αντίστοιχο. Ε, όταν μιλάμε για συγκεκριμένη δράση, νομίζω ότι δεν θα μας βοηθήσει μόνο αυτό. Χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς και ξεκίνησε η εκστρατεία έγκαιρα, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στα πολιτικά κόμματα να διαλέξουν ε, τους καταλόγους των υποψηφίων. Κάθε δεύτερο όνομα, για παράδειγμα, να είναι ένα όνομα γυναίκας. Και θέλαμε να επηρεάσουμε και τα πολιτικά κόμματα, γιατί αυτά είναι αυτά τα οποία ορίζουν και αποφασίζουν ποιοι εν τέλει θα είναι υποψήφοι για να τους ψηφίσουμε. Ε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που άλλαξε την κατάσταση κάποια στιγμή ε, στην δικιά μου τη χώρα ήταν ένα γυναικείο κόμμα. Ε, και νομίζω ότι αυτό φόβησε το πολιτικό κατεστημένο σε τέτοιο βαθμό που ξεκίνησαν μια πιο ενεργή διαδικασία συμμετοχής γυναικών και είχαν και μια πολιτική τέτοιων καταλόγων που σήμαινε ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση γυναικών. Και φυσικά υπήρχε και η απειλή της νομοθεσίας. ήταν ένα είδος σιωπηλή ποσόστοσης αν θέλετε και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο ενθάρρυνε την ίδια την αλλαγή και βοήθησε και τη συζήτηση επί του θέματος στη Σουηδία και αυτή τη στιγμή όλα τα πολιτικά κόμματα εφαρμόζουν την αρχή της ισότητας των φύλων. Δεν θα βρείτε κανένα ηγέτη κόμματος που να σας πει ότι ε, Αυτό η νοοτροπία. Όλοι ε, δραστηριοποιούνται ενεργά για την ισότητα των φύλων, γι' αυτό και έχουμε και υψηλή εκπροσώπηση. Το ίδιο ισχύει και για τη Φιλανδία και για την Νορβηγία. Εγώ πιστεύω στις ποσοστώσεις, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη άλλωστε, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα τρόπο να διορθώσουμε μια υφιστάμενη ανισορροπία και αδικία για μένα είναι ένα πρακτικό εργαλείο, αλλά χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία και χρειαζόμαστε να λάβουμε αποφάσεις και να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Και αυτό είναι σημαντικό και για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες. Αυτό που θα μπορούσε να απαντήσει βέβαια κάποιος και δεν ξέρω κατά πόσον συνέβη αυτό στην Σουηδία είναι ότι ε, ανησυχούμε και για τα σχόλια πίσω από την πλάτη σας όταν μπείτε σε ένα σύστημα λόγω ποσοστώσεων. Μήπως υπονομεύεται η θέση των γυναικών. Είναι καλύτερο να έχετε ένα σύστημα όμως όπου οι άνδρες επιλέγουν άνδρες. Είναι μεγαλύτερο προσόν αυτό. Όταν ε, γυναίκες με προσόντα χάνονται στην αφάνεια. Αυτό είναι το σύστημα που έχουμε σήμερα και ουσιαστικά οι άνδρες επιλέγουν άλλους άνδρες. Δεν το βρίσκω λοιπόν πιο δημοκρατικό ή πιο νομότυπο αυτό. Θα μπορούσε ίσως να είναι πρόβλημα εάν υπήρχε μια κατάσταση όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουμε αρκετέ γυναίκε με προσόντα. Αλλά σήμερα έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε αρκετέ γυναίκε με προσόντα για να πληρώσουν αυτέ τι θέσει. Και εκεί έρχεται και η δημοκρατική πρόκληση για όλου μα και καθήκον μα από εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ, Μάργκοτ. Μήπως θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια παρατήρηση, αλλιώς ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε, η Μάργκοτ μπορεί να μείνει ή να φύγει, ανάλογα με το τι ακριβώς έχει να κάνει σήμερα το απόγευμα. Να ακούσω την παρουσίασή σας πρώτα, να πω πριν ξεκινήσουμε ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, στο οποίο φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκαν για να έχουν μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τις γυναίκες και το ρόλο τους στις εκλογές. Ε, γίνονται όλο και περισσότερες τέτοιες κοινέ προσπάθειες, κυρίως ε, γνωμοδοτήσεις της ε, δημοσκοπήσεις συγγνώμη, του Ευρωβαρομέτρου πέρα από τις ε, τυποποιημένες. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε τώρα και θα ήθελα να ζητήσω από τους δύο ανθρώπους που ασχολήθηκαν με αυτό να έρθουν εδώ και να μας σχολιάσουν τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου και τη Σούζαν Παντίτσι από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ έκανε και μία ανάλυση για μία σειρά από τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου. Uh, Έχουμε λοιπόν την Κλόντια και τη Φίνκα Ντεκούλιν από την Κάλοπ. Πάρε και το καρτελάκι σου. Μπορείτε να κάτσετε όπου θέλετε. Είμαστε ευέλικτες ως γυναίκες. Να ζητήσω λοιπόν ε, από τις κυρίες από την TNS και την Gallup να μας ε, πούνε εντάχει ποια ήταν τα αποτελέσματα, τι μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε, τι διαπιστώσατε και τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτά τα στοιχεία και από εκεί και πέρα η Σούζαν θα μπορούσε να μας πάει λίγο περαιτέρω και να συζητήσουμε βάσει των όσων θα μας πείτε. Κλόντια λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Είναι προνόμιο προφανώς να σας παρουσιάσουμε κάποια από τα αποτελέσματα για την έρευνα που κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, το Κοινοβούλιο ως μια κοινή προσπάθεια όπως επεσήμενε η κυρία Βάλστρομ και αν ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα ε, δεδομένα μπορούμε να τα κοιτάξουμε από τη γυναικεία σκοπιά. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες δεδομένα, εμείς φέραμε ελάχιστα σήμερα και ελπίζω ότι οι βασικές πτυχές θα διαφανούν από όλα αυτά και θα ε, να τα αντιληφθεί και το κοινό μας σήμερα. Το Ευρωβαρόμετρο όπως ίσως ξέρετε, για να σας δώσω και κάποια στοιχεία, είναι μία ποσοτική έρευνα που δίνει ε, κάποια στοιχεία, ένα αντι, αντιπροσωπευτικό δείγμα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεσσάρων υποψηφίων χωρών και λαμβάνει υπόψη της και ένα ευρύ φάσμα ηλικιών από 15 ετών και άνω και γίνεται μεγάλη συνέντευξη γύρω στη μία ώρα με όσους απαντούν και καλύπτεται ένα μεγάλο φάσμα απαντήσεων. Σήμερα επιλέξαμε για σας μία σειρά από τις βασικές πτυχές οι οποίες σχετίζονται με τις εκλογές και με το τι ενδιαφέρει τους ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό περνάει κυρίω σήμερα, ότι το πλαίσιο στο οποίο δίνεται μια απάντηση είναι εξίσου σημαντικό με την ίδια την απάντηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να περάσουμε ως μήνυμα σήμερα δίνοντάς σας αυτή τη συνολική εικόνα. Να σας ε, δώσω ένα περίγραμμα του τι θα κάνω, κάποια πράγματα ως περιεχόμενο που σας είπα ήδη, ποια θέματα επηρεάζουν τις γυναίκες περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες, διότι αυτό ήταν ε, ε, ο σκοπός του νευροβαρομέτρου, να δούμε ε, σε σχέση με πέρσι μια αντιπαρεθεση ανδρών γυναικών και να δούμε τι θα προκύψει για την κατάσταση της ζωής του καθενός και τη μελλοντική προοπτική. Τι είναι το πιο βασικό, διότι για τις γυναίκες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το ερμηνεύσουμε. Δεν είναι η πολιτική αυτή αυτή, αλλά τα καθημερινά θέματα και νομίζω ότι οι γυναίκες που μίλησαν πριν από μένα ήδη επεσήμαναν πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές δυσκολίες που έχουν οι γυναίκες ε, επειδή φροντίζουν και για το σπίτι και γιατί ασχολούνται περισσότερο και με τους άλλους. Ε, βέβαια δεν είναι πάντα ο κανόνας, αλλά ισχύει οι γυναίκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική κοιτάμε μια στενότερη σχέση και από εκεί και πέρα κοιτάμε τις εκλογές ε, και ε, με λίγο στενότερη οπτική γωνία και από εκεί και πέρα έχουμε τα αποτελέσματα. Ως προς το περιεχόμενο τώρα η οικονομική κάμψη δυστυχώς ε, ε, επηρεάζει τους πάντες και το βλέπουμε και από τις απαντήσεις των γυναικών. Σε όλο το ευρωβαρόμετρο μπορούμε να δούμε και τις γραμμές των τάσεων που είναι και ομορφιά των ε, στοιχείων αυτών και βλέπουμε πώς άλλαξε η κατάσταση από το 2007 που είχαμε τα πρώτα στοιχεία της κρίσης μέχρι το φθινόπωρο του 2000 δηλαδή τη σύγκριση 2007 και 2008 που βλέπουμε ότι έχει διαφανεί πλέον η κρίση και βλέπουμε τι δεδομένα έχουμε εκεί. Οι εκλογές δεν είναι και το πρώτο στοιχείο στο μυαλό των πολιτών, αλλά είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα λάβουν υπόψη τους επόμενα, ε, στους επόμενους μήνες. Και έγινε Νομίζω και η σχετική παρατήρηση από την Αντιπρόεδρο, την κυρία Κράτσα, ότι η ανεργία, η οικονομική ανάπτυξη και η αγοραστική δύναμη είναι όλα αλληλένδετα και ε, κυριαρχούν στο μυαλό των γυναικών. Ως προς την εθνική διάσταση, ε, διότι όλα αυτά τα πράγματα, κυρίως η ανεργία ε, επηρεάζει και την οικογενειακή αιστεία και επομένω ε, και εδώ ε, είναι αλληλένδετα τα πράγματα και οι γυναίκες τείνουν να μην απαντούν σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ξέρουν ε, νομίζουμε ότι είναι περισσότερο ειλικρινείς ή πιο διακριτικές όταν απαντούν. Ε, προτιμούν να πούν ότι δεν ξέρουν ε, παρά να υπερβάλλουν σε μία απάντηση. Αυτή είναι μία υπόθεση την οποία λαμβάνουμε υπόψη στα δεδομένα. Δεν έχουμε βέβαια καμία στατιστική απόδειξη από αυτού. Να δείτε τώρα κάποια από τα στοιχεία. Αν δούμε λίγο το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται οι γυναίκες ε, και οι άνδρες, ε, η απεσιοδοξία είναι πιο μεγάλη στις γυναίκες. Ε, όταν βλέπουμε την οικονομία της χώρας ή την κατάσταση απασχόλησης, βλέπετε ότι είναι μια κοινή ανησυχία. Το 66% των ανδρών λένε ότι είναι κακό, αλλά οι γυναίκες ε, ε, είναι σε υψηλότερες. Το ίδιο συμβαίνει και για την ανεργία και από εκεί και πέρα για τις ε, τιμές που αυξάνονται και τον πληθωρισμό. Αυτά νομίζω και η αγοραστική δύναμη την ανέφερα λίγο πριν. Η βασική ανησυχία για μια χώρα είναι τα θέματα αυτά, η οικονομία, το 30% το υποστηρίζουν οι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι 39%. Από τις 28.000 ε, ε, συνεντεύξεις που κάναμε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μεγάλα ποσοστά. Το κατά πόσον αυτά ε, επηρεάζουν τον καθένα προσωπικά, βλέπετε ότι το θέμα είναι να κυριαρχεί περισσότερο στις γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και όταν Ρωτούμε για την οικονομική κατάσταση της οικογενειακής αιστείας ε, και πάλι ε, οι γυναίκες βλέποντας την κατάσταση το τώρα, οι γυναίκες θεωρούν ότι η κατάσταση είναι κακή ή θα χειροτερεύσει. Για τα προηγούμενα πέντε χρόνια οι γυναίκες είναι λιγότερο επικριτικές ε, σε σχέση με τους άνδρες και για το μέλλον είναι το αντίστροφο. Οι γυναίκες είναι πιο ανήσυχες, οι άνδρες λιγότερο. Τώρα, το θέμα του να υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να πληρώνονται οι λογαριασμοί, ε, οι γυναίκες ανησυχούν και πάλι περισσότερο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι η πολιτική δεν είναι το κυρίαρχο θέμα. Ε, δεν τους ρωτήσαμε αν τους ενδιαφέρουν τα επαγγέλματα ή τα αθλητικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά η πολιτική δεν είναι το πρώτο θέμα που συζητούν. Τώρα, για το κατά πόσο οι πολίτες νιώθουν ότι είναι ενημερωμένοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το αν γνωρίζουν ε, απτά στοιχεία. Περίπου το 50% των ανδρών λένε ή ισχυρίζονται ότι ξέρουν πώς ε, λειτουργεί η ισχυριζονται οτι ξερουν πως Ένωση. Οι γυναίκες είναι πιο επιφυλακτικές. Ε, ε, το 36% επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει τα στοιχεία και πάλι βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό. Ε, τώρα, για αυτά στοιχεία ζητήσαμε τέσσερα στοιχεία αν είναι σωστά ή λάθος οι άντρες ήταν πολύ πιο σίγουροι για τις γνώσεις τους και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, όντως εδώ η γνώση φαίνεται ότι ε, γνωρίζουν οι άντρες περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για, στην ερώτηση για το κατά πόσο γνωρίζουν κάτι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή έχουν διαβάσει κάτι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και πάλι βλέπουμε αυτό το κενό. Ε, οι γυναίκες βέβαια τείνουν να μην διαβάζουν τα ίδια μέσα ενημέρωσης με τους άνδρες. Υπάρχει μια λογική, αλλά νομίζω ότι αυτό που περνάει είναι ότι οι γυναίκες λένε ότι παρακολουθούν και επακρυπνούν λιγότερο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ε, τα τρία τέταρτα του γυναικείου πληθυσμού λένε ότι γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δραστηριότητές τους. Εγώ ω ερευνήτρια εδώ θα μπορούσα να σας πω ότι εδώ ανοίγονται κάποιες δυνατότητες. Να μην το θεωρήσουμε δηλαδή ως αρνητικό στοιχείο, αλλά ως μια δυνατότητα που θα μπορούσαμε να απτύξουμε περαιτέρω. Οι γυναίκε επίση έχουν χαμηλότερο επίπεδο στην πεποίθηση ότι ακούγεται η άποψή του. και για τα στοιχεία ως προς την ανεργία, ε, για τη χώρα μου, τι πλήττει το ίδιο με το σπιτικό. Ε, οι γυναίκες τείνουν να ε, συμφωνούν περισσότερο ότι τους ανησυχούν αυτά τα στοιχεία. Τώρα, για το κατά πόσο εισακούγονται οι φωνές τους, η ανησυχία φαίνεται να, να είναι η ίδια και υπάρχει μεγαλύτερη πτώση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες γυναίκες ε, λένε ότι συμφωνούν σε αυτό το στοιχείο. Τώρα για τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν οι εθνικές κυβερνήσεις υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία τους επηρεάζουν ε, περισσότερο στο σπίτι, στην οικογένεια, στην καθημερινή τους ζωή, τους ενδιαφέρει προστασία των καταναλωτών και για τα παιδιά τους, ε, θέματα μεταφοράς, υποστήριξη σε περιφέρειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Και εδώ βέβαια έρχεται και το θέμα της ανεργίας που είναι συνδεδεμένο με αυτό. Τώρα, γυναίκες και πολιτική. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίγο χειρότερη για τις ε, γυναίκες από ότι για τους άνδρες, αλλά είναι πολύ ε, υψηλότερο το ποσοστό των ουδέτερων ε, γυναικών και δεν είναι περισσότερο αρνητικέ από τις γυναίκες. Επομένως το ποτήρι εδώ είναι μισογεμάτο. Και εκφράζονται και κάποιες απόψεις. Τώρα, το κατά πόσο υπάρχουν ωφέλη με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες και πάλι είναι πιο επικριτικές και όσον αφορά την υποστήριξη στο ευρώ, η υποστήριξη των γυναικών είναι πολύ μικρότερη. Και πάλι ε, αυτό έχει σχέση με το γεγονός ότι ε, η αγοραστική δύναμη δεν θεωρήθηκε ότι ευνοήθηκε λόγω του ευρώ. Τώρα, η αξιοπιστία προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι παρόμοια περίπου με τους άνδρες. Φαίνεται βέβαια να μην είναι ακριβώς η τάση ε, να εμπιστευθούν τα όργανα και έχουμε πολύ περισσότερες απαντήσεις δεν ξέρω. Οι γυναίκες φαίνεται δηλαδή να μην ξέρουν τι να πούνε εδώ. Μία στις πέντε γυναίκες απάντησε δεν ξέρω. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ε, σε γενικό βαθμό είναι χαμηλότερη από ότι η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω ότι είναι μια στις πεντε γυναικες απαντησε δεν ξερω εμπιστοσυνη στην κυβερνηση σε γενικο κοβαθμο ειναι χαμηλοτερη απο οτι η εμπιστοσυνη στην ευρωπαικη ενωση αυτο νομιζω οτι ειναι μια εκκληση για να λάβει δράση η ε, εθνική κυβέρνηση και όσον αφορά στις δημόσιες ε, δραστηριότητες, οι γυναίκες και οι άνδρες φαίνεται να συμφωνούν εδώ. Δηλαδή, θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν περισσότερο, που είναι πιο κοντά σε αυτούς, ε, φαίνεται να τους ενδιαφέρουν περισσότερο να τους ενδιαφέρουν και προκύπτει αυτό από τις δημοσκοπήσεις. Τέλος, να δούμε λίγο και τις ε, ψηφοφορίες που είναι εξίσου σημαντικές. Έχουμε τα τρία βασικά θέματα, γιατί θα τα αναφέρω εδώ, η αύξηση των τιμών, η οικονομική κατάσταση και η υγειονομική περίθαλψη. Ε, είδατε νωρίτερα ότι η προστασία των καταναλωτών έχει να κάνει και με την ε, υγειονομική περίθαλψη. Αυτό αφορά την ίδια την οικογένεια λοιπόν και προκύπτει εδώ. Οι βασικές πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βελτίωση της οικονομικής, την της ε, προστασίας των καταναλωτών, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ε, και ε, αυτό έχει να κάνει και με την αίσθηση της ασφάλειας. Και τα τρία βασικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ έχουμε ουσιαστικά τα ίδια πράγματα που είδαμε και πριν. Ανεργία, οικονομική ανάπτυξη και αγοραστική δύναμη. Ε, φαίνεται λοιπόν να ε, επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία και τι ημερομηνίε των εκλογών, μπορεί να μην σα εκπλήξει ή να σα εκπλήξει το γεγονό ότι το 3 τέταρτο των γυναικών δεν ξέρουν πότε θα γίνουν οι ευρωεκλογέ. Ίσως αυτό να αλλάξει όταν θα πλησιάζουμε προς εκλογές. Το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι μικρότερο στις γυναίκες και η πρόθεση ψήφου εδώ ευθυγραμμίζεται και πάλι η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει λοιπόν η απάντηση των γεγονών με το ότι δεν έχω σχέση με την πολιτική, αλλά έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ πρώτα. Η πρόθεση ψήφου λοιπόν, παρά το γεγονός ότι είναι μόνο στο 1 τρίτο, ε, είναι κοινή με τους άνδρες και τα ε, ποσοστά του δεν ξέρω εδώ είναι αρκετά χαμηλά, επομένως φαίνεται ότι δεν ε, αδιαφορούν οι γυναίκες. Όπως σας είπα, ε, οι γυναίκες αγωνιούν περισσότερο και η πολιτική δεν φαίνεται να είναι το κυρίαρχο θέμα στις γυναίκες. Τους ενδιαφέρουν περισσότερο θέματα οικονομίας και που είναι πιο κοντά στην οικογένειά τους και στο σπίτι τους. Και ως προς τη γνώση για τις εκλογές διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, υψηλά ποσοστά μηδενικών γνώσεων και ως προς την πρόθεση ψήφου ε, οι γυναίκες και οι άνδρες φαίνεται να έχουν το ίδιο ενδιαφέρον. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για μια εξαιρετική δυνατότητα να κάνουμε κάποια πράγματα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ, Κλώδια. Θα ήθελα να μας παρουσιάσει τη δική σου άποψη από την Καλόπ. So, well, um, σας ευχαριστώ. Η Κλώδια αναφέρθηκε στο στάνταρτ ευρωβαρόμετρο και μια σειρά δημοσκοπήσεων που έγιναν. Αλλά όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έγινε και μια πολύ ειδική έρευνα που είχε ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξεταστώ συγκεκριμένα οι στάσεις των γυναικών σε σχέση με τις ευρωεκλογές. και σε σχέση με τι δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η έρευνα για την οποία θα συζητήσουμε τώρα. Ορισμένα από τα στοιχεία που θέλω να τονίσω αναφέρθηκαν ήδη. Θα ε, προσθέσω λοιπόν κάποια αριθμητικά στοιχεία. Αυτά θα σας πω. Η έρευνα αυτή έγινε το Φεβρουάριο, έγινε τηλεφωνικά, οι περισσότερε ε, έγιναν με σταθερά, σταθερά τηλέφωνα, ορισμένα όμως και από κινητά και επίσης κατευθείαν σε άμεση άποψη. Ε, ήρθαμε σε επαφή με άντρες και με γυναίκες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αλλιώς τις θέσεις των γυναικών. Εξάζουμε πρώτα λοιπόν την συμπεριφορά για τις εκλογές. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες βασίζουν την απόφασή τους σε θέματα των, ε, <clears throat> της εκστρατείας μετά όσον αφορά το κόμμα και μετά όσον αφορά την προσωπικότητα των υποψηφίων. Βλέπετε ότι οι άντρες περισσότερο συγκρίνουν τα θέματα και όχι τόσο τις προσωπικότητες ως οι γυναίκες. Άμα εξετάσουμε τότε συγκεκριμένα τις εκλογέ για, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι γυναίκες εξετάζουν περισσότερο τα θέματα εμπειρία των υποψηφίων σε ευρωπαϊκά θέματα και όχι τόσο στην πολιτικό προσανατολισμό. Οι άντρε λίγο πολύ το ίδιο βάρο δίνουν και στα δύο αυτά θέματα. Όταν εξετάσουμε τώρα το θέμα της εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό το θίξαμε ήδη σήμερα, αλλά πάνω από το ίμιση των Ευρωπαίων γυναικών αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται σωστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και 4% αισθάνονται πολύ καλά εκπροσωπούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το ίμιση των Ευρωπαίων γυναικών θέλουν 50% και πάνω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου να είναι γυναίκες, ενώ αυτή την ίδια επιθυμία έχουν 39% των ανδρών θέλουν περισσότερε γυναίκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. το εξεταστεί το θέμα που μπορεί να επιτευχθεί αυτό, ελέγχθη σήμερα το η η θελοντική δεσμεύση του κομμάτων, αυτό δεν έτυχε ιδιαίτερη ε, υποστήριξη. Οι γυναίκες δεν θέλουν έτσι θεσμοσυμημένες μεθόδους. Το 27% των γυναικών υποστήριξαν τις ποσοστώσεις, αλλά μόνο 23% των γυναικών οι γυναίκες θέλουν κυρίως να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες για να ασχοληθούν με την πολιτική, όχι τίποτα περισσότερο από αυτό. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τις επόμενες ευρωεκλογές, για να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει την ε, ισότητα των φίλων στην ε, οικογενική ζωή, θα ήθελαν οι γυναίκες να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απασχολούν με παιδιά ή να υπάρχουν πολιτικές που αναφέρονται στη σημασία των ε, νευροφυσικών σταθμών και άλλων σταθμών για τη διατηρήση των παιδιών. Και βέβαια αυτό έτυχε τη υποστήριξη κυρίως των τεωρών γυναικών. Επίσης, οι γυναίκες είπανε ότι το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει την, ε, την εξίσου αντιπροσώπηση των παιδιών από τους δύο γονείς σε περίπτωση διαζυγίου. Κοινή δηλαδή και δαιμονία. Επίσης να προωθηθούν ε, πολιτικές για την ε, ίση αμοιβή και να εξεταστούν ιδιαίτερα θέματα κατά της βίας, κατά των γυναικών και το εμπόριο των γυναικών. οι γυναίκες ε, κυρίως ενδιαφέρονται για ίσες ευκαιρίες απασχόληση και τόσο ίσως για την, ε, τους ίσους μισθούς. Για να ανακεφαλέσω αυτά που είπα, έχω να σας πω ότι γενικά στις, εκλογέ θέλουν οι γυναίκες κυρίως να εξετάσουν τα θέματα που, ε, που συζητούνται και όχι τόσο την προσωπικότητα του υποψηφίου. Όσον αφορά την ίση εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται ότι οι γυναίκες δεν θέλουν τόσο όσο οι άντρες να υποστηρίξουν άμεσα μέτρα και όσον αφορά τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου είπα ότι οι γυναίκες θα ήθελαν να εξεταστεί το θέμα ότι ο χρόνος που ασχολούνται με τα παιδιά τους να ληφθεί υπόψη σαν χρόνος εργασίας αναγνώριση της σημασίας των ε, διάφορων σταθμών για τα παιδιά και ε, ισότητα στην κοινωνία γενικά και θα ήθελαν οι γυναίκες να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ίσους μισθούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Φιούγκα. Θα επανέλθουμε σε κάποια από αυτά τα θέματα σε λίγο γιατί νομίζω θίγησαν κάποια σημαντικά θέματα. Πρώτο το κάνουμε όμως θα ήθελα να ζητήσω από την Σούζαν Μπαντούτσο Επνέξτα να μας παρουσιάσει τη δική της ανάλυση γιατί νομίζω ότι εξετάσετε τρία, τρεις έρευνες και πού καταλήγετε όσον αφορά την στάση των γυναικών και πώς εμπνέονται οι γυναίκες ε, όταν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ή να δεσμευτούν πολιτικά. ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν είναι ένας κόσμος ανδρικός μόνο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία εδώ που υπήρχαν από την Ευρωμερόμετρο και βέβαια τα τελευταία στοιχεία που από την έκτακτη αυτή έρευνα. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν, ε, σε μια παλιά έρευνα θεωρήθηκε ότι η Ευρώπη είναι καλά νέα για τις ε, γυναίκες και ότι εκπροσωπούνται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι εθνικά επίπεδα και επίσης ε, ε, δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι μια, ένας νέος θεσμός σε σχέση με, τα εθνικά κοινοβούλια και γι' αυτό οι δομές είναι πολύ καλύτερες ε, για τις γενίκες, υπάρχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες για τη συμμετοχή τους, είναι ένα όργανο δηλαδή φιλικό προς τις γυναίκες. Και επίσης για δεν υπάρχει επίσημα ένα κόμμα αντιπολίτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί είπαν ότι αυτό είναι ε, προς όφελος των γυναικών. Και όσον αφορά τις πολιτικές και τις νομοθεσίες που εθετούν, ε, υπάρχει γενική συμφωνία ότι πολλές πολιτικές είναι προς όφελος των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όσον αφορά την έκτακτη αυτή έρευνα που παρουσιάστηκε, υπήρχε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το 40% τουλάχιστον των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υψηλό ή έστω και μέση επίπτωση στην ευμάρεια, στην παιδεία, στην πρόνοια και στα δικαιώματα των γυναικών. Και μία πλειοψηφία των γυναικών στην Ελλανδία λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ιδιαίτερε επιπτώσεις αυτούς του τομείς της ζωής τους. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, η ερώτηση αφορά την προσωπική ζωή του απαντώντος, της απαντούσας στις ερωτήσεις. Δεν είναι τα γενικά, αλλά όσον αφορά την εκάστοτε προσωπική ζωή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Αυτό κινεί την έρευνά μου, που είναι η δεύτερη μου παρουσίαση, είναι υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι οι γυναίκες και το πολιτικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοηθεί η πολιτική δέσμευση των γυναικών. Τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο καταδεικνύουν ότι και οι άντρες και οι γυναίκες συμφωνούν ότι οι, της πολιτικής ε, επικρατούν οι άντρες. 71% των ανδρών και το 77% των γυναικών συμφωνούν. Το 80% των γυναικών και το 86% των ανδρών συμφωνούν ότι οι γυναίκες θα έδιναν μια, νέα, μια διαφορετική προοπτική στην πολιτική. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι οι γυναίκες θα ενδιαφερθούν περισσότερο για την πολιτική αν ζουν σε ένα πολιτικό περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες έχουν πολιτικά αξιώματα. Η ορατότητα λοιπόν των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Το τρίτο σημείο της ανάλυσης μας αφορούσε τη μεθοδολογία. Ε, κάποιες στοιχεία της ανάλυσης που σας παρουσιάζω είναι από το Ευρωβαρόμετρο 69 του φθινοπόρου του 2008. Πέραν αυτού όμως, η κύρια τεχνική της ανάλυσης είναι να συγκριθούν οι άνδρες με τις γυναίκες μέσω των ερωτήσεων αυτών. Αν δούμε τις ε, διαφορές όμως βλέπουμε ότι δεν εξετάζουμε μόνο διαφορές όσον αφορά το φύλλο του απαντώντος θεωρούμε ότι το φύλλο του απαντώντος οδηγεί σε μια σειρά εμπειριών που έχουν επίδραση βέβαια στις τελικές απαντήσεις. Ε, όταν εξετάζουμε γυναίκες δηλαδή έχουν διαφορετικές εμπειρίες ζωής ε, λόγω των παιδιών όσον αφορά το πόσο ευάλωτες είναι οικονομικά ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αυτό βέβαια οδηγεί σε διαφορετικές απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Τούτου λεχθέντως πολλές από τις διαφορές που βλέπουμε μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να είναι πολύ μικρές. Αλλά αν επιμείνουμε και δούμε διάφορες κατηγορίες κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία. Δηλαδή οι διαφορές είναι πολύ μεγαλύτερες και όταν εξετάσουμε επίσης ξεχωριστά κάθε κράτος μέλος βλέπω ότι υπάρχουν σημαντικότατα κενά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το πρώτο που εξέτασα ήταν την πιθανότητα συμμετοχή σε εκλογές. Και κάτι που αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι ότι υπάρχει λίγη διαφορά. Μικρή διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν εκφράζουν την πιθανότητα να ψηφίσουν. Και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει πολύ μικρή διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάτι που έχει επίδραση σε αυτή την απόφαση είναι διαφορετικά θέματα, δηλαδή η απασχόληση, η ηλικία και η παιδεία. Και αν λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους παράγοντες, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία πια διαφορά. Έστω και η μικρή διαφορά που υπήρχε εξαφανίστηκε. Δηλαδή τα χαμηλότερα επίπεδα παιδείας και η υψηλότερη πιθανότητα να είναι άνεργες είχαν ε, οδηγήσει στο μικρό αποτέλεσμα προηγουμένως. Άμα προκριστάσουμε τώρα το θέμα της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ήταν ερώτημα του Ευρωβαρομέτρου 69 Άντρες και γυναίκες θεωρούν ότι είναι καλό να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη τους. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ έχουμε γυναίκες που εκφράζουν υψηλότερη πιθανότητα να συμφωνήσουν. Αλλά άμα κοιτάξουμε εδώ τις διαφορές στην έκφραση διαφέροντος στις ευρωεκλογές, και ακριβώς αυτή είναι η ανάλυση από το Ευρωμένο από το είναι ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ άνδρων και γυναικών. Μεγαλύτερη διαφορά εδώ από ό,τι προηγουμένως και έκανα την ίδια ανάλυση, δηλαδή ε, ηλικία, επίπεδα παιδείας και απασχόληση σαν σταθερές. Και βλέπουμε εδώ βλέπετε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανθρώπων και γυναικών όσον αφορά το ενδιαφέρον για τις ε, εκλογές. Λοιπόν, δεν μπορούμε έτσι να εξηγήσουμε τη διαφορά ενδιαφέροντος για τις εκλογές. Και, όπως βλέπουμε πάλι, όσον αφορά τις πιο ευάλωτες ε, ομάδες του πληθυσμού οικονομικά, οι οποίες έχουν ακόμα χαμηλότερο επίπεδο ενδιαφέροντος για τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι διαφορές μεταξύ άνδρων και γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν. Αυτές οι μεταβλητές, δηλαδή η ηλικία, απασχόληση και παιδεία δεν μας βοηθούν να καταλάβουμε γιατί είναι λιγότερο το ενδιαφέρον των γυναικών στις εκλογές. Ακόμα και αν ελέγξουμε το θέμα της υποστήριξης της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι δεν βρίσκουμε μία λύση. Γιατί εξακολουθεί λοιπόν να υφίσταται αυτή η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά το ενδιαφέρον του για την προεκλογική εκστρατεία. Για να επανέλθουμε στο προηγούμενο σημείο, να πούμε ότι το πολιτικό περιβάλλον οδηγεί σε κάποιες διαφορές, θα έλεγα ότι η εκπροσώπηση και η ορατότητα των γυναικών στην πολιτική αρένα είναι αυτό που ε, κάνει τη διαφορά. Εάν οι γυναίκες ήταν πιο ορατές, ή εκεί που είναι οι γυναίκες πιο ορατές, θα ενδιαφέρονται περισσότερο οι γυναίκες. Αυτό που έκανα λοιπόν είναι να εξτάσω αυτές τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε σχέση με το ενδιαφέρον του στην εκλογική εκστρατεία και να δω πώς υπάρχουν εδώ διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών μελών για να το συσχετήσω με την εκπροσώπηση γυναικών από τις χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει μια θετική σχέση. Σας δείχνω εδώ μια σχέση 5 ετών μεταξύ δύο μεταβλητών. Εδώ πρόκειται για μια απλή εικόνα και βλέπουμε ότι εκεί που είναι πιο υψηλή η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική, οι γυναίκε ενδιαφέρονται περισσότερο για τι ευρωεκλογέ. Αν υπάρχουν δηλαδή πολλέ ευρωβουλευτέ ε, γυναίκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυξάνεται το ενδιαφέρον των γυναικών για τι εκλογέ αυτές. Και το κενό αυτό δεν είναι θέμα μόνο ενδιαφέροντος. Γιατί αναφερθήκαμε προηγουμένω και στο θέμα των πολιτικών γνώσεων και τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και όπω είπε η προλαλή σα, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι γυναίκε τι είναι περισσότερο να πούνε, δεν ξέρω. όσον αφορά ουσιαστικέ ερωτήσει. και φανταζ... καταλαβαίνετε ότι αν η ερώτηση είναι σωστό ή όχι οι άντρε, ακόμα και αν μόνο ο, μαντεύουν οι πιθανότητε η απάντηση να είναι σωστή είναι περισσότερος παρά τις γυναίκες που λένε δεν ξέρω όπως το βλέπετε και εδώ. Το ίδιο ισχύει και όταν ρωτούνται για την ημερομηνία των ευρωεκλογέ. Αλλά το κενό μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά το δεν ξέρω σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών μειώνεται το κενό αυτό στις χώρες που αυξάνει το ποσοστό γυναικών ευρωβουλευτών. Πάλι βλέπουμε εδώ να υπάρχει μια απάντηση. Δεν ξέρω. Όσον αφορά πολιτικές γνώσεις σε σχέση με τις ευρωεκλογέ. Ένας άλλος τομέας στον οποίο η εκπροσώπηση των γυναικών παίζει ένα σημαντικό ρόλο είναι όσον αφορά τη στάση εναντί των θεσμικών οργάνων. Και αυτό που έκανε είναι ότι προσπάθησα να δω τι γίνεται με αυτέ τι ερωτήσει εμπιστοσύνη που είδατε προηγουμένω. Έχουν εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι γυναίκε, Φερρυπίν. Πάλι ήταν η ιδέα όταν υψηλότερο το ποσοστό εκπροσώπησης θα αυξηθεί και η εμπιστοσύνη. Το σύγκρινα εγώ αυτό. Γιατί ξέρουμε υπάρχουν σημαντικέ ε, διαφορέ μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά γενικά την εμπιστοσύνη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που έγινε εδώ είναι ότι οι γυναίκε τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο την Ευρω... Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν οι γυναίκες εκπροσωπούν καλύτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, όσο αφορά το ενδιαφέρον για τις εκλογές, γνώσεις για τις εκλογές και στάσεις όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, μπορεί πραγματικά να συσχετιστούν άμεσα όσον αφορά τη μεγαλύτερη ορατότητα των γυναικών. Αν επανέλθουμε τώρα στις ευρωεκλογές του 2004, είναι σημαντικό να δούμε ποιοι θα μπορούσαν να ήταν οι μηχανισμοί μέσα των οποίων οι μηχανισμοί των γυναικών, της ε, συμπεριφοράς των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επιπτώσει στη συμπεριφορά των γυναικών γενικά. Θα επανέλθω τώρα στις εκλογές του 2004. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσο ορατές ήταν οι γυναίκες υποψήφιες εκλογές αυτές και είδαμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά την ορατότητα των γυναικών υποψηφίων. Αυτό που σας δείχνω εδώ είναι το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων σε κάθε κράτος μέλος σε σχέση με το ποσοστό των γυναικών που ακούγονται στα νέα. Και βλέπετε ότι σε ορισμένε χώρε όπω η Αυστρία, η Γαλλία και το Βέλγιο Υπάρχουν σημαντικότερε διαφορές όσον αφορά το ποσοστό των υποψηφίων γυναικών σε σχέση με την κάλυψη από τα ΜΜΕ. Παρόλο λοιπόν που στις χώρες αυτές υπήρχαν πολλές υποψήφοι, η ορατότητά του στα ΜΜΕ ήταν χαμηλή. Και κατά εμέ η ορατότητα στα ΜΜΕ των γυναικών θα ήταν ένας από τους μηχανισμούς μέσα των οποίων οι γυναίκες θα ενδιαφερθούν και θα ασχοληθούν με την εκστρατεία. και μπορούμε έτσι να δούμε πώς άλλαξαν οι απόψει των γυναικών έναντι των ευρωεκλογών κατά τη διάρκεια της εκδρατείας. Αυτό που είδα είναι ότι υπήρχε ε, σημαντική αύξηση όσον αφορά το ότι οι γυναίκες αισθάνονται υπεύθυνε έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίπτωση στην οποία ήταν πιο ορατές οι γυναίκες υποψήφοι. Δηλαδή εδώ βλέπετε όταν είναι ορατές οι γυναίκες υποψήφιες υπάρχει αύξηση της υποστήριξης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτός δηλαδή από θέμα ε, πολιτικής είναι ότι η εκπροσώπηση των γυναικών έχει επιπτώσεις σημαντικές στην συμπεριφορά. Συμπερασματικά. Σε κατακλείδη, μέσα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών και της συμβολική ισχύω που έχουν ε, στην πολιτική, αυτό μας δίνει μία απάντηση του γιατί η πολιτική δέσμευση των γυναικών είναι χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Γιατί η πολιτική δεν θεωρείται ένας κόσμος γυναικείος, εκτός αν οι γυναίκες είναι ορατές και εκπροσωπούμενες. Όσον αφορά το έκτακτο στο ευρωβουλευτικό, ξέρουμε ότι το 70% των γυναικών θέλουν τουλάχιστον 40% γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει αυτή η βούληση δηλαδή για την εκπροσώπηση των γυναικών. Αλλά πώ θα φτάσουμε εκεί, στην αύξηση δηλαδή της εκπροσώπησης των γυναικών, στο ευρωμαρόμετρο φαίνεται ότι υπάρχει μια υποστήριξη πλειοψηφία για την ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετάσχουν περισσότερο. 53% των γυναικών και το 42% των ανδρών θεωρούν ότι αυτή η υποστήριξη είναι αυτό που θα είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν χαμηλά επίπεδα όμως υποστήριξη για τις ποσοστώσεις. 5% και 12% των ανδρών θεωρούν ότι αυτό θα ήταν μια απάντηση θετική όσον αφορά ένα άλλο ερώτημα του εκτάκτου αυτού ευρωβερόμετρου, κατά πόσον θα μπορούσε να ε, ζητήσει το Κοινοβούλιο να έχει περισσότερε γυναίκε στη διαδικασία λήξη αποφάσεων. Μόνο το 5% των γυναικών συμφώνησαν με αυτό και το 8% των γυναικών είπαν ότι αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ότι δηλαδή θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο να τοποθετήσει περισσότερε γυναίκε σε μια διαδικασία λήψη απασχόληση για να βελτιώσει την ισότητα των φύλων. Ε, ακόμα δηλαδή και αν υπάρχει υποστήριξη για την πρόσθεση των γυναικών στη πολιτική, υπάρχει υψηλό επίπεδο υποστήριξης για τις ποσοστώσεις. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν. Ελέγχθη ότι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικός για την πρόθεση των γυναικών και την εκλογή τους. Κόμματα που έχουν σε ηγετική θέση γυναίκες πιο εύκολα θα προωθήσουν γυναίκες σαν υποψήφοι και αν τις προωθήσουν ως υποψήφιες τόσο πιο μεγάλη συμμετοχή να εκλεγούν. Όσον αφορά τους κανόνες για τις ποσοστώσεις είναι επίσης σημαντικές, ιδίως εάν η κουλτούρα ε, του κόμματος ή της χώρας δεν είναι φιλική για την υποψηφιότητα Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ποσοστό είναι πάρα πολύ σημαντικές. Περαιτέρω. Η κάλυψη από τα ΜΜΕ των προεκλογικής εκστρατείας. Άλλο ένα στοιχείο αυτό. Ξέρουμε ότι οι ευρωεκλογές δεν καλύπτονται πάρα πολύ από τα ΜΜΕ. Εκτός αυτού η περισσότερη κάλυψη των ευρωεκλογών έχει σαν στόχο εσωτερικούς ε, πολιτικούς ε, ε, παράγοντες και πάνω σε εθνικά θέματα και όχι ευρωπαϊκό θέματα. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι ότι οι γυναίκες περισσότερο από οι άντρες τείνουν να αποφασίσουν την τελευταία μήνα της εξαρτίας, 55% των γυναικών το είπαν αυτό, ενώ 50% μόνο των ανδρών. Και όπως είδαμε προηγουμένως, ε, θεωρούν ότι τα θέματα της εκτατές είναι πάρα πολύ σημαντικά και βάσει αυτών αποφασίζουν. Γι' αυτό ξέρουμε ότι η περίοδος της προεδρικής εξαρτίας είναι πάρα πολύ σημαντική για τις γυναίκες και αν δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη από τα ΜΜΕ δεν θα έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους που χρειάζονται για να πάρουν αποφάσεις. Για άλλη μια φορά λοιπόν, τα ΜΜΕ και η κάλυψη από το ΜΜΕ είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Αναφέρθηκε το θέμα των ποσοστώσεων. Υπάρχει μια πρόταση για πανευρωπαϊκούς εκλογικούς καταλόγους και αν χρησιμοποιούν ποσοστώσεις πάνω σε αυτό και ιδίως το λεγόμενο zipping, δηλαδή αν να υπάρχει σειρά άνδρας γυναίκα, άνδρας γυναίκα, άνδρας γυναίκα για... όλα αυτά θα αυξήσουν την οραματικότητα και θα βοηθήσουν να εκλογούν οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ καλή ανάλυση, προκαλεί πολλές ερωτήσεις και μου δόθηκε εντύπωση ότι οι γυναίκες εμφανίστηκαν λιγότερο για τις εκλογές, ενώ στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και το ίδιο ε, ισχύει και για την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει κάτι ε, και για τα πολιτικά κόμματα και θα ήθελα να ακούσω και από εσά. Τι συμπέρασμα βγάζετε από όλα αυτά, ε, την αρχική σας αντίδραση. Θέλει κάποιος να κάνει κάποια παρατήρηση ή να κάνει κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή. Ή θα μπορούσα να θέσω εγώ κάποια ερώτηση, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία είναι το τι μπορούμε να κάνουμε με το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μικρή υποστήριξη με την ιδέα των ποσοστώσεων και θεσμικών μηχανισμών για τη λύση του θέματος αυτού. Και έχει σημασία τα πολιτικά κόμματα ε, προχωρούν ε, χωρίς, ε, χωρίς εμάς. Γιατί ουσιαστικά εσύ, Σούζαν, μας λέτε ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της εκπροσώπησης των γυναικών και της συμμετοχής και παρουσίας των γυναικών. Είναι μήπως αυτό κάποιο μήνυμα ε, ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να προχωρήσουν, να προωθήσουν το θέμα των ποσοστώσεων. Θα μπορούσες να μας πεις ε, κάποια πράγματα εσύ ε, ως μέλος του Εργατικού Κόμματος που ετοιμάζει να ξεκινήσει την προεκλογική σου εκστρατεία. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, διότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορούμε να έχετε περισσότερες γυναίκες εκπροσώπους αν έχετε ποσοστώσεις. Από την προσωπική μου πείρα στο Εργατικό Κόμμα, δεδομένου ότι και το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι λίγο διαφορετικό από την υπόλοιπη Ευρώπη, τη στιγμή βεβαιωθήκαμε ότι θα έχουμε γυναίκε στα ψηφοδέλτια, μόνο τότε τι είχαμε στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το παραγράψουμε αυτό. Ω πολιτικά κόμματα θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και να την τηρήσουμε κιόλα. Ε, ελπι... Ήλπιζα να ήταν εδώ η Μάργκοτ, διότι υπάρχουν χώρες στι οποίε υπήρξαν ποσοστώσει και το προχώρησαν το θέμα αυτά και αυτή τη στιγμή έχουν ίση εκπροσώπηση γυναικών, εκεί δεν τίθεται πλέον θέμα ποσοστώσεων. Ε, δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να το συνεχίσουμε και να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει. Έχεις δίκιο, υπάρχουν κάποιες χώρες ε, οι οποίες ξεκίνησαν με τις ποσοστώσεις και τώρα έχουν ε, ισότητα λίγο πολύ. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό νομίζετε. Είναι γι' αυτό που λέγαμε πριν ότι οι γυναίκες ε, φοβούνται ίσως κάπως ε, με την ιδέα ότι ε, μπορεί να έχουν προωθηθεί άδικα. Νομίζω ότι είναι πολλαπλές οι απαντήσεις η ερώτηση δεν ήταν ε, απευθείας ε, υποστηρίζεται ή όχι τις ε, ποσοστώσεις, ήταν θεωρείται κατά πόσον θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός για να ενθαρρύνεται τη συμμετοχή των γυναικών. Λοιπόν, και είναι εύκολη η ερώτηση, απάντηση συγγνώμη, το να μην δεσμευτεί κάποιο με κάτι όπω οι ποσοστώσει. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των γενικών και δεν θα ήμασταν πιο συγκεκριμένοι. Αν λοιπόν η ερώτηση ήταν ε, είστε υπέρ ή κατά των ποσοστώσεων, μπορεί να είχαν περισσότερη υποστήριξη ποσοστώσει. Και ξέρω ότι μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τι ποσοστώσει υπάρχουν γυναίκες υποψήφιες και γυναίκες ε, ευρωβουλευτές που είναι υπέρ των, ε, των ποσοστώσεων. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα του να πούν οι γυναίκες ότι οι ε, ποσοστώσεις θα επιβεβαιώσουν τις διαφορές ε, μεταξύ των φύλων και, ε, και τίθεται τέτοιο θέμα γενικώ. Και το άλλο θέμα είναι ότι αν μιλάμε για πολιτική συμμετοχή, δέσμευση, οτιδήποτε είναι αυτό, διότι ο όρος αυτός είναι λίγο περίεργος, αν κάποιος ως κόμμα, πολιτικό μπορεί να πει έχει σημασία αν ε, το μόνο θέμα είναι αν γνωρίζουν την ημερομηνία για τις εκλογές ή αν νομίζουν ότι ξέρουν κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μας νοιάζει αν οι γυναίκες ε, ασχολούνται με το θέμα αυτό. Κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Αλλά μία από τις κυριότερες εκστρατείες ήταν να πείσουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν στις εκλογές. Φαίνεται ότι αυτό ήταν αρκετά σοβαρό θέμα, τουλάχιστον σε σχέση με τους άντρες. Ίσως ένα από τα θέματα που για μένα προσωπικά και αυτή είναι η προσωπική μου δήλωση, ε, είναι ότι θεωρώ ότι οι ποσοστώσεις είναι διάκριση για να επιτύχουμε ένα στόχο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αναφέρθηκε αρκετές φορές ο όρος, πιο πολύ αφορά το αν θα το προάγουμε και υπάρχει και ερώτηση που έθεσες εσύ. Έχει σημασία. Επειδή εγώ συμμετείχα σε αυτή την έρευνα και διαπιστώνω ότι αυτό που ίσως οι γυναίκες θα θεωρούσαν πιο θετικό ως προς τη συμμετοχή τους είναι να είναι κάτι πιο απτό. Αν οι πολιτικοί και λαποτηλητικά θέματα είναι πιο απτά σε σχέση με την καθημερινότητά τους, και αν δούμε και τα θέματα τα οποία ανακύπτουν και αφορούν την ευμάρεια του καθενός, την οικογενειακή ευμάρεια, αυτή τη στιγμή αυτά γίνονται πιο απτά και δεν ε, είναι τόσο απομακρυσμένα από το οικογενειακό μέτωπο, υπάρχουν πολύ περισσότερες ε, δυνατότητες να συμμετέχει κάποιος. Και μπορεί να ακούγεται πιο συναισθηματικό ως τεχνική, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι ε, το ίδιο τακτικό και λογικό με τους άνδρες. Είναι αλήθεια αυτό, διότι αν δείτε τα στοιχεία θα δείτε ότι είναι από στατιστικής πλευράς ε, σημαντικά για τους καθημερινούς ανθρώπους που δεν είναι στατιστικοί ε, έχουν σημασία. Αν δείτε, για παράδειγμα, το ενδιαφέρον για την πολιτική μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν εγώ ετοίμαζα μία εκστρατεία, θα θεωρούσα ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να υπάρξουν κάποιες πολιτικές οι οποίες θα στρέφονται κυρίως προς τις γυναίκες και όχι στους άνδρες γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο μόνος τομέας στον οποίο φαίνεται να υπάρχει ε, κάποιος σύνδεσμος είναι αυτό το θέμα της εκπροσώπησης και του ενδιαφέροντος. Ιδάλλως δεν φαίνεται να είναι τόσο εντυπωσιακή η διαφορά. Φέμκα, εσύ τι άποψη γι' αυτό. Ω προ την πολιτική, γιατί είμαστε ειλικρινεί εδώ, υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάθε φορά το θέμα που προκύπτει, διότι έχουμε μια σειρά από αριθμού, δείχνουμε διάφορους αριθμού. και ε, σε το θέμα είναι σε ποιο σημείο φαίνεται να έχουν διαφορά αυτοί οι αριθμοί για, τη, για αυτούς που κάνουν πολιτική και το πώς επεξεργάζεται κάποιος τους αριθμούς του είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Ακόμα και αν ε, κάποιες διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες, εξακολουθούν να είναι διαφορές και αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και να μην τα παραβλέψουμε και να πούμε ότι εντάξει μικροδιαφορές είναι. Επιτρέψτε μου να απαντήσω κι εγώ. Ο τρόπος που παρουσιάσαμε τα δεδομένα είναι μια συνολική εικόνα όλων των ευρωπαϊκών χωρών από κοινού. Και αυτό δείχνει κάποιες πολύ προφανείς και πολύ σημαντικές αλλαγές μεταξύ ανδρών και γενικών ε, στα κράτη-μέλη. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, και αυτό το βλέπουμε και αμέσως όταν εξετάζουμε την έκθεση. Και αυτό ήταν και αυτό που σας πρότεινα. Να δούμε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους σε κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερα κενά μεταξύ ανδρών και, τα, και γυναικών, η εκπροσώπηση των γυναικών είναι μία από τις ε, αιτιολογήσεις η οποία ενδιαφέρει εμένα. Δηλαδή λέτε ότι σε κάποιους πολιτικούς τομείς υπάρχουν μεγάλα κενά μεταξύ του τι θέλουν οι άνδρες και οι γυναίκες στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή τα, ο μέσο όρο των στοιχείων μπορεί να μην φαίνεται τόσο εντυπωσιακά. Αν κάνουμε ένα καταμερισμό ανά χώρα μπορεί να υπάρχει διαφορά. Όντω, σε κάποια από τα κράτη-μέλη ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η ανεργία και τα οικονομικά θέματα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη τριάδα όλων των χωρών. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές ε, τεράστιες διαφορές μεταξύ αυτών, αλλά ε, το ευρωβαρόμετρο ε, είναι τόσο μεγάλη έρευνα που έχει τη δυνατότητα να μας δώσει όλα τα στοιχεία ανά χώρα και όντως υπάρχουν διαφορές στα άλλα θέματα, στα ίσονα σημασία θέματα που προκύπτουν και θεωρείτε ότι αυτό έχουν να κάνουν και με τα θέματα ανακράτος μέλος. Δεν έχουμε κάνει την ανάλυση αυτή τη στιγμή μεταξύ φίλων και σε επίπεδο χώρας, γιατί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν εστιάσαμε σε αυτό και νομίζω ότι ούτε η Γκάλοπ εστίασε σε αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πιο εντυπωσιακέ διαφορές. Ε, για παράδειγμα, το έγκλημα σε κάποιες χώρες μπορεί να είναι πιο ε, σημαντικό για τις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Ενώ σε επίπεδο ε, όλων των χωρών να είναι σε κατώτερη κλίμακα. Βάσει της συγκεκριμένη αυτής έρευνας εξετάσαμε πώς διαφέρουν οι άνδρες και οι γυναίκες και πώς είναι οι διαφορές ανά μέλος. Συνήθως έχουμε ένα παρόμοιο ε, μοντέλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν διαφορές και υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες είχαμε την αντίθετη τάση στις χώρες μέλη. Και οι χώρες διαφέρουν μεταξύ τους και ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πάντα ο αντιπροσωπευτικός αριθμό για τις χώρες. Ένα από τα σχόλια που έγιναν είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, προβάλλονται οι γυναίκες υποψήφιες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχει να κάνει με το ποιο φαίνεται στις ειδήσει και ποιο όχι. Ε, κάποιος από τους δημοσιογράφους ίσως ε, στο κοινό έχει άποψη από αυτού. Εμένα προσωπικά με κατέπληξε αυτό, διότι ε, διαπιστώνω ότι πολλές από τις γυναίκες υποψήφιες είναι πιο ενδιαφέρουσες από τους άνδρες. Ε, εμείς βάζουμε περισσότερες γυναίκες ε, στο πρόγραμμά μας, αλλά φαίνεται ότι εγώ είμαι μειοψηφία. Ως δημοσιογράφος πάντα του λένε ή το ρωτάνε από τα ευρωπαϊκά όργανα να περάσει και ένα μήνυμα. Και Το μήνυμα δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά οι πληροφορίες είναι σίγουρα το σημαντικό κομμάτι. Έχετε καμιά ιδέα λοιπόν για το πού θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αν διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο σε σχέση με όλες τις εκλογές. Είμαι από την Ουγγαρία, Βικτόρια Σούς. Εργάζομαι για ένα φεμινιστικό περιοδικό και υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των γυναικών πολιτικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και των ανδρών. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό στην Ουγγαρία, αλλά οι γυναίκες πολιτικοί πολλές φορές παρουσιάζονται με βάση των ρούχων που φοράνε ε, ή των παραδοσιακών τους ρόλων. Τι καλές σύζυγοι που είναι, αν μαγειρεύουν καλά και πώς είναι η εξωτερική τους εικόνα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλαδή τείνουν να μην εστιάζουν σε αυτά που λένε, που λένε αλλά στο πόσο θηλυκές είναι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα πολιτικό να παρουσιάσω οποιοδήποτε θέμα, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν εστιάζουν στο μήνυμα αυτό καθεαυτό, αλλά στο πώς φαίνεται μια γυναίκα. Και έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο στο οποίο προσπάθησα να κάνω μία σύγκριση ε, για το πώς ε, παρουσιάζονται οι γυναίκες και οι άνδρες πολιτικοί. Η εικόνα είναι τελείως διαφορετική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν εστιάζουν ποτέ ε, απλά και μόνο στην εικόνα μιας γυναίκας. Χάθηκε το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Δεν ακούγεστε, πατήστε το μικρό κουμπάκι δίπλα σας. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο πολύ πέρασε το μήνυμά σας. Ίσως εδώ θα έπρεπε να ρωτήσουμε τους έξι, νομίζω έξι μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουμε, δημοσιογράφους ε, και ανθρώπους του τύπου. Θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε εδώ στο Προεδρείο, αν έχετε να, προσθέσετε οτιδήποτε οι τρεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και νομίζω ότι ε, θα σας ακούσουμε και στο μέλλον. Έχουμε βάλει τα μπελάκια, επομένως ε, μπορείτε να βρείτε το καρτελάκι με το όνομά σας και να καθίσετε. Έχουμε έξι γυναίκες εγνωσμένου κύρου στο κλάδο τους. Tricks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 ομιλία με τους έξι παρισταμένους και θα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένη νομοθεσία λίγο μετά από αυτό για να δούμε πώς περνάει, ε, τι, ποια πράγματα είναι υπαπτυμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας παρουσιάσω λίγο τους ομιλητές μας, την Άντζελα Μπουτιλιόν εδώ εξ αριστερών μου. Θα μπορούσατε να βρείτε λίγο περισσότερα στα μικρά στοιχεία που σας έχουμε δώσει. Είστε από την Ιταλία, από την ε, ΡΑΗ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η Μπέατριξ Κάμπελ είναι πολύ γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα άρθρα της και για τις ε, μεταδόσεις της. Είστε και μέλος των Πρασίνων, οπότε μπορείτε να μας εκδηλώσετε ανοιχτά το πολιτικό σας ενδιαφέρον και είστε μέλος και της Εθνικής Επιτροπής ε, Γυναικών. Δίπλα σας είναι η Ειρήνη Καρανασοπούλου. Είστε και εσείς δημοσιογράφος από το 1986 και ειδικεύεστε σε ευρωπαϊκά θέματα και διπλωματικά θέματα και έχετε και μία κόρη 12 ετών όπως και εγώ. Δίπλα σας η Πιλάρ Μαρτίν από το Ισπανικό Δημόσιο Ραδιόφωνο, διευθύντρια του Ραδιοφώνου 1. Εδώ στα δεξιά μου η Άντζελα Μίλ από το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, διευθύντρια του European Publishers Council και δίπλα είναι η Mercedes Hindereg από το Bavarian Hunt Food και είστε διευθύντρια αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού. Νομίζω ότι όλες σας θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα πράγματα για πέντε λεπτάκια, να μας πείτε για κάποια πράγματα που ακούσετε και να μας πείτε λίγο και την προσωπική σας πείρα ε, για το πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι σας επηρέασαν ή ε, επηρεάζονται οι γυναίκες ε, στις χώρες σας από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τι νομίζετε ότι περιμένουν οι πολίτες από τις ευρωεκλογέ, κυρίως οι γυναίκες. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, να ξεκινήσουμε από δεξιά και να συνεχίσουμε. Μερσέντες. Yes, um, I will start and I will start in... Θα ξεκινήσω, θα μιλήσω γερμανικά. Μετά συζήτηση θα περάσω πάλι στα αγγλικά, αλλά για την πρώτη μου παρουσίαση να σας τα πω γερμανικά. Εδώ και 30 χρόνια είμαι ε, δημοσιογράφος και είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να αρχίσω με πολιτική δημοσιογραφία, γιατί με ενδιαφέρει αυτό, αλλά στην αρχή της δεκαετίας του 70 στη Γερμανία υπήρχαν πολύ λίγες γυναίκες στην πολιτική δημοσιογραφία, ειδήσει, σχόλια κλπ. Και όταν εγώ παρόλα αυτά πήγα σε μια πολιτική ένδυμαση σαν ελεύθερη επαγγελματίας, μου είπαν ότι μπορώ να τα γράψω ό,τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να παρουσιάζω τι συμβολέ μου, γιατί δεν είναι αρκετά σοβαρέ οι φωνέ των γυναικών να παρουσιάσουν πολιτικά θέματα. Και πράγματι τότε εγώ ήμουνα μόνη γυναίκα μεταξύ πολλών ανδρών. Εγώ ένα ελεύθερη επαγγελματία, οι άλλοι είχαν μόνιμη θέση απασχόληση. Όταν προσπάθησα να μονιμοποιηθώ κι εγώ, ήταν αδύνατον σε αυτό το πρόγραμμα ειδήσεων και θα μπορούσα μονάχα να μονιμοποιηθώ στο πρόγραμμα για την νεολαία. Και ο επιφοκαφαλής προσωπικού με ρώτησε τότε το θέλεις πράγματι γιατί δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες από εκεί και Δηλαδή θα μπορούσα να παραμείνω στο πρόγραμμα για τα παιδιά ή των γυναικών. Εγώ δεν το συζήτησα το θέμα, είπα βλέπουμε. Ε, εργάστηκα στο πρόβλημα αυτό για την ολέα και μετά έγινε κάτι άλλο, δηλαδή ε, απόκτησα οικογένεια, έχω και μια κόρη 27 χρονών σήμερα και δεν ήθελα να εργάζομαι πλήρη απασχόληση. Τότε για δημοσιογράφους ήταν αδύνατο, σε εμά τουλάχιστον. Ήταν δυνατό αυτό για τις γραμματείς, ήταν δυνατό για το τεχνικό προσωπικό αλλά όχι για τις δημοσιογράφους. Και γι' αυτό καταρχήν έφυγα από την ε, ε, ραδιοφωνία και πήγα ως ε, υπεύθυνη της Γερμανικής Σχολής Δημοσιογραφίας. Το 1995 έγινα επικεφαλής εκεί ήταν επαναστατικό στη Γερμανία, δεν υπήρχε καμία ε, διευθύντρια δημοσιογραφικών σχολών γιατί ο προσαρμοσμός ήταν στο, στους κύριους δημοσιογράφους των ε, μεγάλων εφημερίδων και αυτοί είναι και ήταν και είναι άντρες. Δεν θέλω να απτύξω τα πάντα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για αριθμικά στοιχεία αν σας ενδιαφέρει. Εγώ θα ήθελα στη συζήτησή μας καταρχήν να ακούσουμε πού υπάρχουν γυναίκες δημοσιογράφοι γιατί στην πολιτική μόνο το 15% είναι γυναίκες ενώ γενικά τουλάχιστον στη Γερμανία είναι κάθε τρίτος δημοσιογράφος γυναίκα. η εικόνα ανδρών και γυναικών πώς προωθείται στα ΜΜΕ. Η συνάδελφος από την Ουγγαρία είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε και αυτό να το συζητήσουμε, δηλαδή πώς παρουσιάζονται όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες. Και για τι πράγματα ενδιαφέρονται οι γυναίκες όταν χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, τι διαβάζουν, τι ακούνε, τι βλέπουν. Ε, ακούνε περισσότερο ραδιόφωνο και βλέπουν περισσότερη τηλεόραση από τους άνδρες ε, διαβάζουν λιγότερες εφημερίδες, τουλάχιστον στη Γερμανία. Αυτό ίσως σχετίστηκε με το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες δημοσιογράφοι που γράφουν στις εφημερίδες αυτές. Εξεπλάγει όταν ε, άκουσα τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων ότι άντρες και γυναίκες ενδιαφέρονται εξίσου για την πολιτική. Δημοσκοπήσεις στη Γερμανία δεν απέδεσαν αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. Για τους άντρες είναι περισσότερο πολιτική, αθλητισμός, τεχνολογία, ενώ άλλα θέματα, οικογένεια, περιβάλλον, μόδα, είναι θέματα που διαφέρουν τις γυναίκες. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε νομίζω. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα των γυναικών όταν χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ. Έτσι, το προτείνω αυτό. Σαν μια ερώτηση για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι αυτό οδηγεί στο εξή. Αν καλύπτεται για παράδειγμα, την προεκλογική εκστρατεία για τι ευρωεκλογέ, πώ θα το καλύψετε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ενδιαφέρον. Ε, για μένα είναι μια μεγάλη πρόκληση, είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα και για το ίδιο το κοινοβούλιο άλλωστε. Πώ ε, μπορεί να περάσει την νομοθεσία. Άντζελα, θα μπορούσα να σου ζητήσω να μα δώσει μια εικόνα του πώ ήταν τα πράγματα για σένα στη Βρετανία για να φτάσει μέχρι εδώ που έφτασε και κατά πόσον ενδιαφέρει για αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, ότι ένας μεγάλος αριθμός γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει σε πολιτικές που είναι φιλικές προς τις γυναίκες και κατά πόσον αυτό εκτιμάται ή είναι γνωστό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω από κάτι το οποίο με διασκέδασε στην αρχή όταν μιλούσατε με τη Μάργκοτ Βόλστρομ την πρώτη φορά που μπόρεσα εγώ να ψηφίσω σε γενικές εκλογές ήταν η πρώτη φορά που ψηφίσαμε ε, μια γυναίκα ε, πρωθυπουργό το 1979. Ό,τι και να πιστεύετε για την πολιτική της Μάργαρετ Θάτσερ δεν ήταν ε, μια συνηθισμένη γυναίκα. Και φυσικά ήταν η πρώτη φορά που είχαμε και άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και η πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν γυναίκα. Ε, από πολύ νωρί λοιπόν οι προσδοκίες μου για αυτά που μπορούσαν να επιτύχουν οι γυναίκες ήταν αρκετά υψηλέ. και ε, είχα και μια τάση προς την πολιτική αλλά τελικά διάλεξα μια διαφορετική κατεύθυνση. Θα σας πω μια προσωπική ιστορία γιατί νομίζω ότι άπτεται λίγο των θεμάτων που ακούσαμε σήμερα. Πέρσι το καλοκαίρι μιλούσα με το 17χρονο γιο, του, γιο μου και την 21 ετών κόρη μου, η οποία είχε προσφάτως ξεκινήσει να δουλεύει, το αφεντικό της είναι γυναίκα και μιλούσαμε για καριέρα, πληρωμές, προοπτικές και εργαζόμενες μητέρες. Και ήταν μια από αυτές τις καθοριστικές στιγμές που δεν την περίμενα και καθόλου. Ως εργαζόμενη μητέρα φανταζόμουν και φοβόμουν πάντα ότι τα παιδιά μου ε, σε κάποια στιγμή θα ένιωθαν άσχημα για το χρόνο που, ε, της απουσίας μου, διότι λόγω της δουλειά μου έκανα και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Και αυτοί έλεγαν στους φίλους τους τι καταπληκτική καριέρα πίστευαν ότι έχω, τι ενδιαφέροντα που είναι όλα αυτά τα ταξίδια και δεν ξέρουν πώς κατάφερα να τους φροντίζω και να φροντίζω και ένα σπιτικό ε, ενώ ταυτόχρονα ασχολιόμαι με τη δουλειά. Ε, μπορώ να σας πω όμως ότι δεν ήταν εύκολο. Όταν τα παιδιά μου ήταν πολύ μικρά, ε, τα υβρεφονικιακοί σταθμοί στη χώρα μου τουλάχιστον ούτε καν είχαν επινοηθεί και ή τέλο πάντων δεν ήταν ε, στις προδιαγραφές που θα θέλετε να είναι και δεν υπήρχε καμία ε, πρόβλεψη στο σχολείο για τα παιδιά. 20 χρόνια αργότερα υπάρχει πολύ περισσότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία και κυβερνητικές παρεμβάσεις και πλέον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι εργαζόμενες γυναίκες έχουν πολλές ε, επιλογές ε, για φροντίδα για τα παιδιά τους, η οποία είναι και εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων και υπάρχουν και οι άδειε μητρότητα ε, ε, και ευέλικτα ωράρια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις ε, εργαζόμενες μητέρε. Αυτοί που, ξέρουν, που με ξέρουν θα ξέρουν ίσως ότι εγώ προσωπικά δεν ήθελα να γίνω εργαζόμενη μητέρα, απλώ έτυχε, το είπα στα παιδιά μου και πραγματικά τα παιδιά δεν με πίστεψαν ε, κοίταξαν ο ένας τον άλλον και άρχισαν να γελάνε και είπαν μα, μα, μα άμα δεν είχες καριέρα δεν θα ήσουν αυτή που είσαι. Και εγώ προσωπικά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι ήμουν ένας άνθρωπος που θα με προσδιορίζει η καριέρα μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά οι γυναίκες έχουν την τάση να μην ενδιαφέρονται. Και ίσως αυτή είναι ένας από τους φραγμούς ε, για να φτάσουμε στην κορυφή. Εργαζόμουν με μερική απασχόληση, ήμουν αυτοαποσχολούμενη μάλιστα όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχα προγραμματίσει. Προέκυψε γιατί δεν είχα κάποια δυνατότητα να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω επαμοιβή και ε, δεν ήταν τόσο φιλικά προς τις γυναίκες τα πράγματα τότε. Θα αφήσω μερικά χρόνια πίσω, αλλά όταν ήμουν στον 7ο μήνα ε, στο δεύτερο μου παιδί ε, και για λόγους που δεν έχω χρόνο τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, με προσκάλεσαν σε μια συνεδρίαση που ήταν ουσιαστικά η ιδρυτική συνεδρίαση του European Publishers Council. με είχαν καλέσει για να παρουσιάσω τον ε, Μέρντοκ ε, στους ομοτήμους του και τα σχέδια του για την Ευρώπη, για τις ε, επιχειρήσει σε, θέματα μέσω μαζικής ενημέρωσης και τις απειλές διαφήμισης. Στο τέλος της συνεδρίασης μου ζήτησαν αν ήμουν διατεθειμένη να ε, διοικήσω αυτόν τον οργανισμό βάσει των όσων του είπα για τις απειλές που υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχε κάποιος οργανισμός, ήταν ουσιαστικά συμβουλευτική δουλειά. Ε, ανατρέχοντας βέβαια στο παρελθόν με δύο μικρά παιδιά, μάλλον ένα μωρό παιδί και ένα το οποίο ε, πρόκειται να γεννηθεί, ε, δεν είχα δικαιώματα, δεν υπήρχαν αυτοαπασχολούμενοι, δεν υπήρχε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δεν υπήρχε πρόγραμμα υγείας ε, ή ούτε επίδομα ενεργείας Αλλά ε, να σας πω ότι εγώ ε, απόλαυσα όλη αυτή τη διαδικασία της αυτοαπασχολούμενης, μου άρεσε που βρέθηκα στις Βρυξέλλες. Και ε, να σας μιλήσω λίγο και για τον οργανισμό μας. Από το 1981 μέχρι σήμερα, από 12 εκτελεστικούς διευθυντής περάσαμε στις 28. Τότε είχαμε, στην αρχή είχαμε μόνο τρεις γυναίκες ε, στο EPC. Οι δύο από αυτές, με περηφάνεια μπορώ να πω, ε, είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι οι μόνες γυναίκες που βρίσκονται σε προεδρικό επίπεδο στον οργανισμό μας αυτή τη στιγμή η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για τις γυναίκες και ελάχιστες γυναίκες φτάνουν σε διοικητικά καθήκοντα και νομίζω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν ε, οι συντάκτες ε, για, τα, για τις πολιτικές, τα πολιτικά θέματα ή τα τρέχοντα γεγονότα συνήθως ε, είναι να τα κάνουν άνδρες. Μπορεί να τα ξέρετε εσείς καλύτερα στη χώρα σας, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες παρουσιάστριες τηλεόρασες, αλλά πίσω από το παρασκήνιο η δύναμη μένει στους άνδρες. Και μετά από 20 χρόνια ε, νομοθεσίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο δεν θεωρώ ότι αυτό είναι έλλειψη νομοθεσίες και φυσικά δεν είναι και λόγω έλλειψης ικανοτήτων από πλευράς γυναικών. Κάπου όμως οι γυναίκες φαίνεται να, να κρατιούνται, να μένουν πίσω. Δεν ξέρω αν είναι επειδή θέλουν να διατηρήσουν αυτή την ισορροπία εργασίας και εργασιακής ζωής και οικογενειακής ή αυτό που κάποιος είπε αυτή την εβδομάδα σε κάποιο έντυπο ότι δεν θυμώνουν αρκετά με τους άνδρες. Δεν ξέρω αν θα το αλλάξει αυτό περισσότερη νομοθεσία. Υπάρχει το μεγάλο χάσμα ε, μισθοδοσίας ακόμα, αλλά μια κάποια ισορροπία κατά τα άλλα φαίνεται να έχει επέλθει. Υπάρχουν και θετικές διακρίσεις στη χώρα μου για γυναίκες ε, βουλευτές και υπάρχει και μια μεγάλη καμπύλη που δείχνει την αύξηση των γυναικών στο θέμα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό αλλάζει και λίγο την ε, οπτική με την οποία βλέπουμε την ε, πολιτική. Δεν είναι πλέον ανδροκρατούμενη. η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζει και ε, θέτει σε ισχύ κάποιες διατάξεις ε, ε, και ούτω καθεξής. Αλλά όλα αυτά είναι και θέμα των γυναικών στο Κοινοβούλιο, γιατί και αυτές ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Όπως ακούσαμε όμως και από την ε, συνάδελφα από την Ουγγαρία, ε, δεν ε, έχει σταματήσει τους άνδρες πολιτικούς και μάλιστα φοβάμαι και κάποιους άνδρες δημοσιογράφους που κάνουν σεξιστικά σχόλια για τα μαλλιά τους, για τα ρούχα τους, για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα οικονομικά και αυτό είναι κάτι το οποίο η νομοθεσία δεν θα μπορέσει ποτέ να αλλάξει. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι άνδρες νιώθουν για τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Δεν θα σου πω ότι η επικεφαλή τη BBC είναι γυναίκα και τη πολιτική πολιτικέ ε, επίση. Άντζελα. Τα θέματα που έδειξε η Άντζελα όσον αφορά τη σημασία τη ε, προδίδα των παιδιών και των προτύπων ρόλου των μοντέλων που όπως είπαμε είχατε εσείς κάτι σας βοήθησε στην καριέρα σας για να φτάσετε εκεί που φτάσετε σήμερα. Είμαι η τρίτη γυναίκα δημοσιογράφος που μιλάει και είμαι η τρίτη που αυτοπροσδιορίζεται από τα παιδιά της. Νομίζω ότι όλες εμείς πριν μιλήσουμε για τη δουλειά μας, για το επάγγελμά μας, μιλήσαμε για τα παιδιά μας. Και Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό και για τη συζήτηση για την πολιτική. Διότι το πρόβλημα των γυναικών στην πολιτική, και εγώ είμαι πεπισμένη από αυτού, είναι ότι οι γυναίκες είναι μητέρες και όλα όσα συνεπάγεται αυτό. Μια γυναίκα είναι ελεύθερη, είναι ελεύθερη να πολεμήσει, να κάνει καριέρα, να ακολουθεί την έμπνευσή της, να ε, χρησιμοποιεί στην ευφυΐα της, όλα αυτά μέχρι ότου γίνει μητέρα. Εκείνη τη στιγμή η ελευθερία της προσδιορίζεται μέσω των παιδιών της. Εάν ε, δεν ε, την βοηθήσουν στη διαχείριση και στην ανάπτυξη των παιδιών, στη διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά της. Μην ξεχνάμε πόσες μητέρες τη σήμερον ημέρα είναι ε, ανήπανδρες μητέρες. Η υπόλοιπη ζωή της λοιπόν, ο όλος αυτοπροσδιορισμός της, ε, πέρα από τον ρόλο της μητέρας, είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Ε, να σας πω ότι εγώ έκανα τέσσερα παιδιά, ε, χάρη και στην τύχη να έχω μια ζωή η οποία έγινε στο εσωτερικό μια επιχείρηση, δεν περιορίστηκε η ελευθερία μου. Έγινα δημοσιογράφος στα 23 μου, κέρδισα, ε, πέρασα κάποιο διαγωνισμό και έγινα δημόσιο υπάλληλο στη ΡΑΗ και ε, η μητρότητά μου ήταν εγγυημένη από ε, συγκεκριμένη νομοθεσία μεγάλη μου κόρη είναι 23 χρονών, η οποία μου επέτρεψε να κάτσω πέντε μήνες στο σπίτι και να φροντίσω το κοριτσάκι μου και μετά βέβαια χρειάστηκε να προσαρμοστώ γιατί και στην Ιταλία τότε δεν υπήρχαν ακόμα βρεφονεπιακοί σταθμοί, αλλά τέλος πάντων υπήρξε η δυνατότητα με κάποιο τρόπο να τη ζήσω αυτή τη μητρότητα. Τα τέσσερα παιδιά βέβαια, όταν μιλάμε για καριέρα, ε, σαφώς επιβράδυναν την καριέρα μου αν κάποιος είναι δημοσιογράφος, είναι απλά δημοσιογράφος. Δεν έχει θέμα καριέρας, είναι δημοσιογράφος, υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες αυτού του επαγγέλματος, γράφει, κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση, κάνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, ε, γράφει σε μια εφημερίδα, ε, είναι ο αγωγός για κάτι άλλο, είναι συντάκτης, πάντα όμως είναι δημοσιογράφος. Ε, μιλάμε όμως πάντα για καριέρα, εγώ αυτή τη στιγμή είναι διευθύντρια που είναι το, η κορυφή της καριέρας του δημοσιογράφου και έλεγα ότι η προσωπική μου ζωή, την οποία δεν στερήθηκα για λόγους πληρότητας της ζωής μου, ε, τη, βήτα, τη ζωή πρέπει να τη ζούμε σε όλες τις, εκφάνσεις. Ε, έλεγα λοιπόν ότι η καριέρα μου επιβραδύνθηκε φυσικά για λόγο ευτυχών συγκυριών ε, και για κάποιες προσωπικές ε, για τη δυνατότητα να διαχειριστώ το χρόνο μου ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας ε, και της δουλειάς και έφτασα τελικά σε αυτό που θεωρείται το top της καριέρας μου. Ε, το 1979 όταν εγώ ξεκίνησα με τις ε, ειδήσει στην τηλεόραση υπήρχε μόνο μία γυναίκα που ασχολούνταν με το θέμα αυτό. Όταν εγώ έγραψα το πρώτο μου άρθρο για τις εκλογές στη Γερμανία ο διευθυντής είπε μια βρισιά και μετά είπε είναι αδύνατο να το έχει γράψει αυτό το άρθρο μια γυναίκα. Δυστυχώς βέβαια γι' αυτό το είχε γράψει μια γυναίκα αρκετά πεισματόρα και έτσι έκανα το πρώτο μου άρθρο και από εκεί και πέρα ξεκίνησα με έναν τρόπο εργασίας που πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήταν πολύ εύκολος, αλλά το λέω σήμερα μετά από 40 χρόνια. Τότε δεν ήθελα να το παραδεχτώ ούτε καν στον εαυτό μου, γιατί θα ήταν παραδοχή της ήττα μου. Ε, ακολούθησα λοιπόν το δρόμο μου, χωρίς ε, να ανησυχώ για τα σχόλια του ενό ή του άλλου. Προχωρούσα, έκανα τη δουλειά μου, η οποία πάντα με πάθιαζε και νομίζω ότι τμήμα της επιτυχίας μου, αν μπορούμε να την καλέσουμε επιτυχία, ε, οφείλεται και στο γεγονός ότι έχω ένα πάθος για αυτή τη δουλειά. Ε, μετά από 40 χρόνια ε, οι δημοσιογράφοι γυναίκες στη χώρα μου είναι οι μισές του συνόλου του δημοσιογραφικού ιταλικού κύκλου. Υπάρχει μια γυναίκα που διευθύνει ε, μία από τις πιο ε, ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά εβδομαδιαία. Υπάρχουν πολλές γυναίκες αρχισυντάκτριες. Πολλές γυναίκες έχουν ε, και καθήκοντα ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Είναι κρίσιμη η μάζα, όπως έλεγε την πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Άλλες όχι. Άλλες, όπως έλεγε ε, και κάποιος εδώ είναι πιο ικανοποιημένες με την παρουσίαση τηλεοπτικών προγραμμάτων ε, και να μην αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία του μοχλού ε, ενός δελτίου ειδήσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι γυναίκε τείνουν να το ξεχνούν κάποιες φορές. Για να έρθω στα γρήγορα στην πολιτική, στη δεκαετία του 70 ε, συζητούσαμε ε, να να μιλάμε για ποσοστώσει για τι γυναίκε, το 80 πάλι για ποσοστώσει για τι γυναίκε. έχουμε φτάσει το 2000 τόσο και ακόμα συζητάμε για ποσοστώσει για τι γυναίκε. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, οι γυναίκε φτάνουν στην πολιτική αν κάνουν πολιτική, αν υπάρχουν στα πολιτικά κόμματα, αν μάχονται εντό των πολιτικών κομμάτων και δεν κάνουν πολιτική στι εκλογέ. Φτάνουμε μέχρι τι εκλογέ. Επομένω, χρειάζεται να γίνει όλη αυτή η προκαταρκτική δουλειά η οποία είναι κουραστική και πολλές φορές και βαρετή, ακόμα και στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων, γιατί εκεί δίνεται η πολιτική μάχη. Εγώ είμαι σχεδόν πεπισμένη, το λέω βέβαια χαμηλόφωνα, ότι οι γυναίκες δεν έχουν διάθεση να κάνουν πολιτική. Και γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί ήθελαν να κάνουν τις δημοσιογράφους, ε, μιλάω για τη χώρα μου, ξέρω πάρα πολύ καλά και κάποιες άλλες χώρες ε, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αν θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι, κάνουν του δημοσιογράφου. Αν θέλουν να κάνουν του δικαστέ, κάνουν του δικαστού. Οι διαγωνισμοί για του δικαστέ άνοιξαν στι γυναίκε το 1960. Σε 50 χρόνια λοιπόν οι γυναίκε είναι άνω των 50% του δικαστικού σώματο τη Ιταλία. Πρόκειται λοιπόν για μια πορεία η οποία είχε κάποιο αποτέλεσμα. Το δεύτερο όμως ε, σημείο που με ανησυχεί περισσότερο σήμερα είναι ότι αυτή τη στιγμή τελείωσε η μεγάλη μάχη για τις ιδεολογίες ε, των αρχών του προηγούμενου αιώνα που αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Στον 21ο αιώνα το φαινόμενο που βλέπω να αναδύεται πολύ ανασυχητικά είναι η αδιαφορία για την πολιτική. Είναι η αδιαφορία των νέων γενεών και αυτό είναι το στοιχείο και σήμερα και το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των ε, συζητήσεων όλων των πιθανών κινήτρων για να προσεγγίσουμε τις νεότερες γενναίες με την ε, πολιτική. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να σας ε, πω την εμπειρία μου και ευχαριστώ όλους όσους με προσκάλεσαν, αλλά είναι μια ιστορία του παρελθόντος η δική μου εμπειρία. Τα προβλήματα που αντιμετώπισα εγώ ε, για τις γυναίκες, οι κόρες μου δεν τις αντιμετώπισαν. Είναι άλλα τα προβλήματα για τις γυναίκες σήμερα και τα άλλα, προβλήματα, τα προβλήματα που οι νέοι, άνδρες και γυναίκες ζητούν από την πολιτική το οποίο βρίσκεται, εγώ πιστεύω, και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ε, στην αναζήτηση μια νέα ταυτότητα για τον ίδιο μα τον εαυτό. Ε, χάθηκαν οι ιδεολογίε κάποιοι όροι που ε, χρησιμοποιούσαμε στην ιστορία, η δεξιά, η αριστερά, αυτή τη στιγμή είναι καινού περιεχομένου. Και επομένω, και εδώ ολοκληρώνω, βρισκόμαστε εν μέσω μια ολόκληρη διαδικασία μεταμόρφωση, στην οποία οι γυναίκε έχουν ένα θεμελιώδη και ουσιαστικό ρόλο, αλλά μόνον εάν το επιθυμούν. Ευχαριστώ, Άντζελα. Πάρα πολύ. Συζητάμε πώς έχουν προχωρήσει οι γυναίκες προσωπικά και πώς χρησιμοποιούν οι γυναίκες τη θέση την οποία και αντιμετωπίζουν τα θέματα των γυναικών. Υπήρχαν ίσως μεγάλα βήματα στον κόσμο των ΜΜΕ, αλλά όπως είπατε αυτό το θέμα της ένδυας εξακολουθεί να υπάρχει, ιδίως για τις γυναίκες. Για πέστε μας, πού φτάσατε εσείς στο δικό σας ταξίδι και πού βλέπετε το ρόλο των γυναικών στα ΜΕ όσον αφορά την πρόοδο, πολιτική δέσμευση κλπ. Εμένα η δημοσιογραφική μου ζωή άρχισε τέλος δεκαετίας του 60. Υπήρχε μία, μία γυναίκα δημοσιογράφος σε εμάς. Συντάξεις για τους, ειδήσεις ήταν ο, ένας που λόγω και αυτό που έλεγε τουλάχιστον πέντε φορές την ημέρα Και σας λέω, μία γυναίκα εκεί ήταν μία γυναίκα που περίσευε κατά κάποιον τρόπο. και πέρασα στην τε... δημοσιογραφία τεχνολογίας και μετά έγινα ρεπόρτερ όπως είμαι από τότε. Είναι ένα παράδοξο. Σίγουρα οι γυναίκες της δικές μου γενιάς, της ε, γενιάς του Women's League, της απελευθέρωσης των γυναικών, ήμασταν τότε νέες, για τις νέες γυναίκες σήμερα η δημοσιογραφία είναι ένα σημαντικός χώρος δράσης και βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ πολιτική δημοσιογραφία, οικονομική δημοσιογραφία, όλα αυτά που θα ήταν κλειστά κάποια στιγμή. Αλλά αυτό είναι και μια εποχή που τροποποιήθηκε όλη η δημοσιογραφία. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ ε, περιττή δημοσιογραφία, εκατομμύρια δέντρων που χρησιμοποιούνται για περιοδικά όπως το ξέρετε. Αυτά που λένε για τους γνωστά τα ονόματα τα διαβάζω και εγώ δεν λέω. Και υπάρχουν βέβαια και σοβαρές εφημερίδες από την άλλη μεριά. Αυτό που θα ήταν δηλαδή σημαντικό, αυτό που ήταν για μένα αν θέλετε, το, ε, άρθρα πολύπλοκα. 2.000, 5.000, 10.000 λέξεις. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Στη χώρα μας δεν είναι πια ο σύνθετος τρόπος εκείνους με τον οποίο αντιμετωπίζουν θέματα. Και το επάγγελμα αυτό προσελκύει εκα... χι... χιλιάδες ε, φοιτητών στη δημοσιογραφία που ποτέ δεν θα μπορέσουν να εργαστούν στον τομέα αυτό. Γιατί έχουμε μία ε, συμπίεση της ε, δημοσιογραφίας έντονη Τη σωστή δημοσιογραφία. σω είναι κάπω υποκλητικό αυτό που σα λέω. Α, θα σας πω δύο λόγια για το πού πιστεύω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πολιτική μας ατζέντα και η Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε μία κρίση για το πώς παρουσιάζουμε το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, για της ε, εικόνα της γυναίκας που γίναμε μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο, μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε και τι θα οδη... βελτίωνε την κατάσταση. Θα σας το πω πολύ ομά. Υπήρχε η ιδέα, καθόλου τη διάρκεια ζωής μου, ότι εμείς είμαστε μία αποτυχία της ε, εξέλιξης της ζωής και έπρεπε να συμμετάσχουμε, να αναπτυχθούμε κλπ. Τα κάνουμε όλα αυτά. Τώρα εξακολουθεί να υπάρχει η εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε μία μακρά αργή εξέλιξη προς κάποιο σημείο σύγκλησης με τους άντρες. Και η ποιότητα ακριβώς των φύλων είναι αυτό που χαρακτηρίζει. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό έχει τελειώσει. Το πρότυπο ποιότητα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ καλό και που τροποποίησε την νομοθεσία για την ισότητα βοήθησε πάρα πολύ. Και ήταν δραματικά σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο η ειρηνευτική διαδικασία οδήγησε όχι μόνο στο τέλος του πολέμου στη Βόρεια Ολλανδία, αλλά την δυνατότητα μιας δραματικά διαφορετικής δημοκρατίας. Μια δέσμευση για την ηθική ισότητα που χαρακτηρίζει όλη την πολιτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό προήρθε από κάποιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η μακρά αργή πορεία έχει τελειώσει τώρα οδήγησε στο ότι η περίοδος της πατριαρχίας ε, λύγει. Σε 25 χρόνια δεν άλλαξαν πολλά πράγματα όμως. Πέρσι η διαφορά μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών de facto αυξήθηκε. Το πιστεύετε αυτό. Μέσα στα πλαίσια μιας κυβέρνησης εργατικής, το, το, η διαφορά αυτή που είχε μείνει σταθερή εδώ και δεκαετίες αυξήθηκε. Υπήρχε μια γενική εντύπωση ότι όταν οι γυναίκες είναι πιο επαγγελματίες, όταν μπουν μαζικά στην αγορά εργασίας θα αλλάξει κάτι δραματικά στις οικογένειες, στην πολιτική κουλτούρα, στις σχέσεις ανδρών και γυναικών και γυναικών και παιδιών κλπ. και Αυτό που είδαμε είναι ότι αυτό δεν είναι αληθές. Ότι οι σχέσεις των ανδρών προς την οικιακή εργασία, προς τη φρονίδα των παιδιών, κατά βάση δεν έχει αλλάξει από την ε, ε, δεκαετία του 70. Ας πούμε, το 1961 την εποχή που σεβόταν κανένα τον πάτερ φαμίλια, οι άντρε κατά μέσο όρο ήταν 6 λεπτά την ημέρα για τη φροντίδα των παιδιών του. Ο πατέρα μου ερχόταν, ερχόταν σπίτι, έπινε το τσάι του, α, άλλαζε, πλενόταν και έβγαινε. Ήταν επισκέψη στην οικογένεια και δεν ήταν ο σίγουρα. Σήμερα ο μέσος ε, πατέρας ε, ασχολείται 16 λεπτά την ημέρα με τη φροντίδα παιδιών του. Και όσον αφορά την οικιακή εργασία, κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα, κατά μέσο όρο. Ε, επειδή έχουμε όμως ε, στην αγορά εργασία μία διαφοροποίηση. Γυναί, ε, αφενός και όλοι από την άλλη. γιατί κατά μέσο όρο οι μητέρες εργάζονται λιγότερες ώρες σε πληρωνόμενη εργασία και πολλές πολλές πολλές ώρες σε μη πληρωνόμενη εργασία, σε μη αμοιβόμενη εργασία. Και από την άλλη μεριά έχουμε τους άντρε που εργάζονται με αμοιβόμενη εργασία τι πιο μακριές ώρες απασχόληση από όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό οι διαφορές αυξάνονται. Και το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι παρόλο που υπήρχαν σημαντικέ μετατροπές τη κυβερνητικής πολιτική τελευταία δεκαετία από μια κυβέρνηση που θεωρείται ότι είναι φιλική προ τι γυναίκε κατά τη γνώμη μου δεν είναι αληθές αυτό, πολλές από τις κινήσεις που έγιναν, έγιναν μόνο όταν κάποια πολιτική που δείχνει να είναι υπέρ των γυναικών συγκλίνει με άλλες αλλαγές και άλλες πολιτικές. Τα καλύτερα που έκανε η Βρετανική κυβέρνηση είναι να εισάγει μια τεράστια διεύρυνση των κέντρων φροντίδας παιδιών είχαμε το πιο χαμηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Οι εργατικοί το έκαναν. Γιατί ε, τοποθετήθηκε υπέρ των παιδιών ή των γυναικών η κυβέρνηση. Όχι, απλώς θέλουν κάπως να σταματήσουν τα παιδιά από το να γίνονται εγκληματίας. Γιατί φταίγανε οι μητέρες βέβαια για την κακή συμπεριφορά των αγοριών τους. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό πλαίσιο με στο οποίο θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πρέπει να είναι η επόμενη επανάσταση φίλων για να είμαστε σίγουρες ότι δεν θα περιοριστούμε στο μέλλον στις μικρές θεσούλες που μας δίνουν σήμερα. Ευχαριστώ θα ακούσουμε κάποιες από τις ιδέες σας που περνάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη Να δώσω το λόγο στην Ειρήνη τώρα, να μας πει κατά πόσον αυτά σας θυμίζουν κάτι, ποια είναι η δική σας κατάσταση. Γιατί εργαζόστε κι εσείς για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ίσως είσαστε πιο εστιασμένοι προς τα θέματα αυτά. Ίσως είμαι κάπως βαρετή μετά από ακούστε την κυρία Κάμπελ. Εμεί θα το κρίνουμε. Uh, Ένα θέμα που είπε η κυρία Κάμπελ ότι ανήκει στη γενιά της ε, Women's League. Εγώ είμαι από εκείνες τους τυχερές ανθρώπους που η μητέρα μου ήταν της γενιάς αυτής. Και εκείνη ήταν τυχερή που ο πατέρας μου ήταν ένας από τα πολύ πολύ σπάνια δείγματα άντρων που ήταν φεμινιστές από μόνοι τους. Πολύ ε, ευτυχές λοιπόν ε, περιβάλλον για μένα. Δεν ξέρω τι πολλές γυναίκες είχαν αυτό του τύπου το ε, περιβάλλον. Ιδίω στην Ελλάδα όπου έχω ζήσει την περισσότερη ζωή μου. Και επειδή υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα μπορώ να είμαι μια ανήπαντρική μητέρα. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια μερική απασχόληση και τέτοια. Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζομαι 12 ώρες την ημέρα και κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με τη μικρή. Και αυτό το ζευγάρι φεμινιστών είναι εκείνο που ασχολείται με το παιδί μου. Πολύ τυχαίρι λοιπόν. Αλλά να σας τα πω από την αρχή, όταν ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου τηλεφωνήσαν για να συμμετάσχω εδώ, μου είπαν ότι ξέρετε έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε αυτές τις καταπληκτικές γυναίκες από τα ΜΜΕ που θα έρθουν είναι όλες διευθύντριες, ε, ψηλό επίπεδο Αλλά στην Ελλάδα εξετάσαμε όλες τις εφημερίδες και δεν βρήκαμε καμία γυναίκα. Πουθενά σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε αναγκασμένοι να σε καλέσουμε σένα. Ε, μα συγχωρείς πολύ, αλλά τι να κάνουμε. Γιατί η επόμενη θέση είναι πολιτικό συντάκτη και πρέπει να σα καλέσουμε σένα που είσαι πιο μεγάλη εφημερίδα. Εγώ είπα, μην ανησυχείτε. Τα ξέρουμε εδώ έχει χρόνια. Ποτέ δεν θα έχουμε γυναίκα διευθύντρια ή αρχισυντάκτη. Ε, αυτά τα ξέρουμε. Το δεχτήκαμε πια, δεν μας απασχολεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι εργαζόμαστε λιγότερο. Μάλιστα το 1993, όταν έγινα πολιτική συνάκτρια, ήμουστα η πρώτη της ομάδας εκεί. Και ήταν ένα τμήμα του παιχνιδιού, γιατί ο τότε διευθυντής της εφημερίδας έχει αποθάρρυνε μεταξύ, είχε βάλει στοίχημα με τον συντάκτη μιας άλλης εφημερίδας της ομάδας ότι μπορεί να έχει μια γυναίκα και θα πετύχει. Ο άλλο είπε όχι, δεν θα πετύχει. Παίζανε δηλαδή. Αλλιώ ποτέ δεν θα είχε συμβεί αυτό. Ένα παιχνίδι μεταξύ ανδρών. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά δεν θα ήθελα να ε, συγκεντρώσω την προσοχή μου στη, στη προσωπική μου ζωή και πώς εργάζομαι εγώ προσωπικά. Απλώς είχα υποσχεθεί στο διευθυντή μου ότι να σας πω ότι σύμφωνα με, με αυτόν το κύριο πρόβλημα στην Ελλάδα, πρέπει να το τονίσω ότι μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν διαφορετικοί διαγωνισμοί για άνδρες ή για γυναίκες. Το πιο μεγάλο πρόβλημα, λέω, για τις ε, γυναίκες δημοσιογράφους είναι ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να συνδυάσουν την εργασία τους με την οικογενειακή του ζωή. Και αυτό τους κάνει πάρα πολύ ενοχλημένα όταν ενθάζονται, σκέφτονται τα παιδιά τους. Όταν είναι με τα παιδιά τους, σκέφτονται τη δουλειά τους. Είναι μεταξύ των δύο δηλαδή και αγωνιούν συνεχώς. Δηλαδή η Ειρήνη αυτό τονίζει ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ακούσουμε σε λίγο και δύο ευρωβουλευτές που εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα για τις οικογένειες και θα δείτε ότι μερικά από αυτά που συζητάνε και που προτείνουν υπάρχουν σε 11-12 χώρε μέλη, αλλά σε άλλες χώρε δεν υπάρχει όμω. Ναι, ναι, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψει. Α πούμε αυτός, ο διευθυντή άλλο διευθυντή. Πει εντάξει Ειρήνη, έχεις μία κόρη 12 χρονών, θα σου επιτρέψει να εργάζεσαι με μερική απασχόληση. Εγώ δεν θα συμφωνούσα, γιατί αυτό θα με έβαζε αμέσως σε μία υποδέστερη θέση σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους. Δηλαδή θα ισχύει για όλους, Δηλαδή, οι άντρε συνάδελφοι δεν ε, απασχολούνται μόνο 16 λεφτά την ημέρα με τα παιδιά του. Όλοι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα ευελιξία ή δεν θα ισχύει για κανέναν. Αλλά όχι πάλι οι κακόμενε οι γυναίκε που έχουν μωρά, του στείλουμε στο σπίτι του. Όχι. Γιατί πάλι θα έχουμε σε μια κατάσταση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ας επανέλθουμε σε αυτό σε δύο λεπτά είναι πιλάρα θα μπορέσει να μας δώσει κάποια ιδέα. Γιατί όταν μιλάω με γυναίκες στην Ισπανία, θυμάμαι είχα πάει στη Γρανάδα, στο Πανεπιστήμιο και κάναμε μια συνέντευξη για τις γυναίκες στην Ισπανία και ο καθηγητής μου είπε, η καθηγήτρια μάλλον μου είπε, ότι θεωρούσε ότι η συμμετοχή της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τεράστια διαφορά για τις γυναίκες, για την κατάσταση αυτό ήταν λόγω της νομοθεσίας, λόγω της αντιμετώπισης, δεν κατάλαβα ακριβώς. Η δική σου άποψη ποια είναι. Εγώ έρχομαι εδώ να, να αναγνωρίσω δημοσίως ότι εγώ είμαι ε, καρπός ε, της ποσόστοσης του 50%. Αν δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή νομοθεσία, δεν ε, το είχε προωθήσει το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν ε, το είχε προχωρήσει και η κυβέρνηση της Ισπανίας, εγώ ποτέ δεν θα είχα γίνει διευθύντρια του Ράδιο 1, που είναι ένα από τα βασικά... Ε, ένας από τους βασικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ισπανίας. Εγώ ε, συμμετείχα σε αυτή την εκπομπή και με ε, προσπερνούσαν όλοι και όλοι φεύγοντας λέγανε αυτή η κοπέλα είναι πολύ καλή και με πρότειναν ε, για να λάβω τη θέση τους. Αλλά κανένας δεν με είχε σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή για πραγματικά να λάβω τη θέση. Το λέω αυτό γιατί εγώ μέχρι κάποια στιγμή ήμουν κατά των ποσοστώσεων, της ποσόστησης του 50% γιατί ε, όχι γιατί θεωρούσα ότι είναι μια θετική διάκριση. Ε, αντίθετα, από ανοησία πίστευα ότι εμείς μπορούμε να έχουμε περισσότερο από αυτό το 50%. Ένιωθα λοιπόν ότι την απορρίπτω αυτή την πρόταση, αλλά ε, παραδέχομαι ότι είναι καρπός αυτής της ποσόστοσης η θέση που κατέχω αυτή τη στιγμή. Η θέση που κατέχω είναι και ε, προπομπός ε, ε, σε πολλά θέματα. Η επιχείρηση στην οποία εργάζομαι είναι μία από τις πρώτες που έδωσε ισότητα σε θέματα εργασίας γυναικών και ανδρών, κυρίως ως προς τα θέματα δικαίου. Δεν ξέρω στην πράξη τι γίνεται. Να πούμε το εξής. Έχουμε τον ίδιο μισθοδοσία, μπορεί ο καθένα να λάβει τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο υπό την προπόθεση ότι έχει τι κατάλληλε επαγγελματικέ δεξιότητε και τα κατάλληλα προσόντα. Και οι αναλογίε στι διάφορε κατηγορίε είναι ισότιμοι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το 80% των ατόμων που θέλουν να δουλέψουν στο δημόσιο τομέα είναι γυναίκε. και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα, θα πρέπει να το αναλύσουμε. Επιλέξαμε αυτόν τον τύπο των επιχειρήσεων γιατί μας εγγυώνται ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επαγγελματική και οικογενειακή ζωή καλύτερα. Ε, έκανα και εγώ δύο παιδιά, εργάζομαι 22 χρόνια σε αυτή την επιχείρηση και δεν είχα πρόβλημα να τα φροντίσω σε συγκεκριμένε χρονικέ περιόδου. Αλλά πάντα υπό την προπόθεση ότι κατέχει τα κατώτερα κλιμάκια, τι κατώτερε βαθμίδε ε, θέσεων. Δηλαδή, σε όλε τι περιπτώσει ε, είσαι σε υποδεώστερη θέση. Όταν μιλάμε για ποσοστά, ίσω να υπάρχουν και περισσότερε γυναίκε στο ραδιόφωνο, στο κρατικό ραδιόφωνο από ότι άνδρε. Αλλά αν δούμε τι μέσε και υψηλότερες θέσεις, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Αν μιλάμε για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έχει περίπου 40 ή 50 προγράμματα, το 1 τρίτο μόνον ε, έχουν διευθυντή μια γυναίκα. Τα 2 τρίτα είναι άνδρες ε, σε μια επιχείρηση στην οποία το 80% περίπου είναι γυναίκες. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση και αυτό ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ζητήσω να ξεκινήσουν και να ενισχυθούν ε, πολιτικές πραγματικής ισότητας. Και συμφωνώ με τις συναδέλφους ότι ε, ορισμένες φορές ε, η εφημερία ε, χάνεται υπέρ της συμφωλίασης. Διότι ε, το θέμα αυτό το δέχονται τελικά μόνο οι γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Εμεί ζητάμε να ισχύει για όλες τις γυναίκες, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και να αφορά όλες τις γυναίκες. Εμένα προσωπικά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ίδια θέση με τις αδέλφους. Αλλιώς ε, χρειάζεται να δουλεύω 14 ώρες τη μέρα, αλλιώς δεν θα είχα το πόστο που έχω αυτή τη στιγμή. Στην Ισπανία βασιζόμαστε πάρα πολύ στην οικογενειακή βοήθεια, στους παππούδες, στους γονείς, ε, διότι αν μια γυναίκα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αφιερώσει αυτές τις 14 ώρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να βρίσκεται για να έχει ένα πόστο σαν αυτό που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, ε, δεν ε, θα έχει τη θέση της. Και πολλές φορές οι άνδρες το επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να μην διορίσουν μια γυναίκα ε, σε αυτό το πόστο είναι γιατί λένε ότι δεν υπάρχει ευελιξία και δεν έχουμε γιατί η κοινωνία μας έχει φορτώσει με μια σειρά από πάρα πολλά κοινωνικά θέματα και συγκεκριμένες οικογενειακές υποχρεώσεις και πρέπει κάπου να σπάσουν όλα αυτά. Δεν λέω ότι θα πρέπει να χάσουμε τις υποχρεώσεις μας που έχουμε ως μητέρες, απλά λέω ότι είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικέ οι οποίε θα μα επιτρέπουν να έχουμε καλύτερα σχολεία, καλύτερου ε, σταθμού για τα παιδιά μα και όταν εργαζόμαστε ε, να μην νιώθουμε ότι εγκαταλείπουμε την οικογένειά μα και όταν είμαστε με την οικογένειά μα να μην νιώθουμε ότι εγκαταλείπουμε τη δουλειά μα. Εγώ γι' αυτό έχω έρθει εδώ, για να διεκδικήσουμε αυτό. Οι γυναίκε πρέπει να συμμετέχουμε περισσότερο και να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά τα αιτήματα είναι δικά μας. Σα το λέω αυτό γιατί ορισμένε φορές στη δουλειά μου όταν βλέπω ότι ένας άνδρας είναι κάνει κάτι το οποίο είναι αντιφεμινιστικό ε, ε, τότε το δέχομαι ενώ αν το έκανε μια γυναίκα θα τη σκότωνα και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω καθημερινά. Πρέπει να εμπλακούμε και εμείς περισσότερο λοιπόν. Όλες αυτές ε, οι αιτήσει θα πρέπει να είναι αιτήματα τα οποία τα πιστεύουμε στην πραγματικότητα και ε, εάν θέλουμε να συμμετέχουμε στην πολιτική θέλουμε πραγματικά το 50% των βουλευτών των χωρών μας ε, να είναι γυναίκες για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια ισότητα και θα υπάρχει και μια κοινωνική ισότητα γιατί αλλιώς υπάρχει δημοκρατική ε, ανισορροπία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ε, μιλήσαμε λίγο ευρύτερα λοιπόν για το τι θέλουν οι γυναίκες, ε, ακούσαμε τις προσωπικές σας μαρτυρίες, ε, κάποιες ιδέες, περάσανε κάποια σαφή μηνύματα για το αυτό που εσείς ως ε, γυναίκες θεωρείτε. Χρειάζεστε περισσότερη προστασία και υποστήριξη, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες. Να περάσουμε τώρα σε πιο συγκεκριμένα πράγματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι κάνει αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να σας ζητήσω να μείνετε και να συμμετέχετε στο επόμενο κομμάτι της συζήτησης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κράτσα από το Κοινοβούλιο και θα τη ζητήσω να κάνει μια εισαγωγή για τους ε, εισηγητές, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ε, υπεύθυνοι για αυτό το οικογενειακό πακέτο. Θα σας εξηγήσει η ίδια γιατί περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για τους ε, αυτοαπασχολούμενους. Αυτό είναι ένα από τα θέματα το οποίο θα προκύψει σε αυτή την ε, νομοθεσία. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την επέκταση των ε, δικαιωμάτων τα οποία ήδη υπάρχουν και σε άλλους. I'm being asked by the gentleman uh, to uh, ask. Ο κύριος μου ζήτησε να σας ζητήσω να πάτε όλες ε, στις θέσεις σας και από εκεί και πέρα μπορείτε να συμμετέχετε κάλλιστα στη συζήτηση. Κυρία Κράτσα, θέλετε να έρχετε στο Προεδρείο. Well, και μπορούν να έρθουν και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθα όπως βλέπετε και με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι μαζί σας το, προς το τέλος αυτής της συζήτησης, η οποία πιστεύω να υπήρξε πλούσια ε, για όλες και για όλους. Ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι του πολιτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είχα την ευκαιρία να πω στην αρχή στο opening αυτής της ε, το Ευρωβαρόμετρο, φαντάζομαι ότι θα είχατε την ευκαιρία να τα αναλύσετε αυτά κατά τη διάρκεια της ειδική ενότητας, ε, μας πληροφορεί ότι οι Ευρωπαίοι δεν, ε, ε, δεν γνωρίζουν αρκετά την, τη σημασία που έχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ζωή των γυναικών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι κλείνουμε αυτή τη συζήτηση, με, αυτή τη συνάντηση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι συνάδελφοι που είναι δεξιά μου η κυρία Στριντ Λούλινγκ από το Λουξεμβούργο, η συνάδελφος κυρία Εστρέλα από την Πορτογαλία, ε, μέλη της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Ευκαιριών ε, θα αναφερθούν σε δύο ε, δραστηριότητες δικές τους στο πλαίσιο του, της πολιτικής μας από, ε, του, και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Και θα κλείσει η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Ζαμπόρσκα, βουλευτής από την Σλοβακία, η οποία θα έλθει στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ανάγκη να γνωρίσουν οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, το ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζοντα τις αρχές της ισότητας και τις πολιτικές που εφαρμόζει για να πετύχουμε το στόχο της ισότητας. Πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ομοθεσία, με τη στρατηγική αλλά και την εφαρμογή της ισότητας σε όλες τις πολιτικές και τις εκφράσεις του Κοινοβουλίου, το οποίο θέλει να είναι ένα πρότυπο θα μου πείτε αυτός είναι ένας στόχος άπιαστος, η προσπάθεια για να γίνει ένα πρότυπο ε, στην εφαρμογή της ισότητας τόσο στις πολιτικές όσο και στη λειτουργία του, στη δομή του, στη διοίκησή του. Θα δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς στην κυρία Λούλινγκ, η οποία κυρία Λούλινγκ, η κυρία Εστρέλα λέει το πρόγραμμά μας. Η κυρία Εστρέλα έχει πρώτα το λόγο, η οποία η κυρία Εστρέλα είναι ε, η ραπορτέρ για μια έκθεση που έχει να κάνει με την ε, ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων εγγύων, αλλά και των γυναικών που πρόσφατα έχουν ε, αποκτήσει παιδί και βρίσκονται σε αυτή την ευαίσθητη φάση. Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε. Ε, thank you very Ευχαριστώ πολύ θα μιλήσω πορτογαλικά, γι' αυτό κρατήστε τα ακουστικά σας. Η παρουσίαση βέβαια είναι στα αγγλικά. Για μένα όμως είναι πιο εύκολα να τα πω στα πορτογαλικά. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Uh, E, como já foi dito pela Presidente da Mesa e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, eu sou a relatora do they said that it will be it will be able δεν υπάρχει διερμηνία από τα πορτογαλικά. But they said to me that it will be the passive interpretation.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 με συγχωρείτε, τα είχα ετοιμάσει στα πορτογαλικά. Σήμερα είμαι πολύ κουρασμένη βέβαια, ήταν μια μεγάλη μέρα για μένα. Και έχω και μια άλλη συνεδρίαση γιατί η ομάδα των σοσιαλιστών ε, έχουν μια συζήτηση για την ισότητα και θα πρέπει να πάω και εκεί. Θα ήταν καλύτερα δηλαδή για μένα να μιλούσα πορτογαλικά, αλλά τι να κάνουμε. Uh, this directive, it's from 85. Αυτή η οδηγία Χρονολογείται από το 1985. Και υιοθετήθηκε σε όλες τις χώρες, μεταφέρθηκε στις χώρες και στόχος είναι να βελτιώσουμε την υγεία και την ε, προστασία σε θέματα ασφαλείας που προσφέρεται σε έγκυες εργαζόμενες ή σε γυναίκες ε, κατά την περίοδο του θυλασμού. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους κοινωνικούς εταίρους, έχει μια συνδυασμένη νομική βάση προστίθεται το άρθρο 141.3 των συνθήκων το οποίο εισαγάγει την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και η προσθήκη αυτή μας επιτρέπει να εισάγουμε και την έννοια της ε, άδεια πατρότητας. Και αυτό είναι και το βασικό θέμα, η βασική πρόταση της έκθεσής μου. Να υπάρχει καταμερισμός των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα κράτη-μέλη Η άδεια μητρότητα κυμαίνεται μεταξύ 14 εβδομάδων Αυτό είναι το ελάχιστο που προτείνεται από την οδηγία, οι 14 εβδομάδες, και φτάνει μέχρι τις 52 εβδομάδες. Αλλά η μισθοδοσία διαφέρει πάρα πολύ μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία κρατούν ε, το μισθό στο ακέραιο, στο 100% και κάποια άλλη τα οποία κάνουν περικοπή του μισθού. Για παράδειγμα, έχετε εδώ ένα κατάλογο κρατών μελών, τα οποία κρατούν το ακέραιο του μισθού, αλλά Υπάρχει διαφορά ως προς τη διάρκεια. Στη Δανία και στη Μάλτα έχουμε 40 εβδομάδες και στην Εστονία έχουμε 20 εβδομάδες. Τώρα εδώ στη διαφάνεια, στα αριστερά έχουμε την πρόταση οδηγίας από το 92. η οποία προτείνει τις 14 εβδομάδες και έχουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είναι 18 εβδομάδες. Η δική μου πρόταση ως εισηγήτρια είναι το ελάχιστο να είναι 20 εβδομάδες. Γιατί προτείνω 20 εβδομάδες. Διότι αν έχουμε ήδη τις 14 εβδομάδες και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι λίγο πολύ 18 εβδομάδες, δεν είναι μεγάλη διαφορά να περάσουμε στις 20. Επομένως πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα να προτείνουμε 20 εβδομάδες. Βεβαίω θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, και δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης. στην οδηγία υπάρχουν υποχρεωτικά δύο εβδομάδες πριν και μετά τον τοκετό στην πρόταση του της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε έξι εβδομάδες μετά τη γέννα και ε, η δική μου πρόταση είναι οκτώ εβδομάδες ε, μετά τη γέννα. Γιατί όπως ξέρετε χρειάζεται κάποιος χρόνος να ανακτήσει δυνάμεις, να συνέλθει κλπ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τα έχω αλλάξει όλα τώρα και δεν έχω... Τα χαρτιά μου είναι στα πορτογαλικά. Θα ελέγξω αν έχω κάτι εδώ. για την ε, πληρωμή. Στην οδηγία προβλέπεται ένα κατάλληλο επίδομα το οποίο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κατώτερο της ε, ε πληρωμής ε, της άδειας ασθενείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πλήρη καταβολή του μισθού και να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση ε, πτώση κάτω ε, της ε, άδεια ασθενεία. Η πρότασή μου είναι 100% της πληρωμής και να μην είμαστε κάτω του 80%. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες δεν θα χάσουν οικονομικώς γιατί αποφάσισαν να κάνουν παιδιά. Και φυσικά υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ξέρω ότι στα διάφορα κράτη-μέλη το ποσοστό για, την, ε, για τις πληρωμές για την αποζημίωση ασθενείας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα, η απαγόρευση απόλυση. Οι αλλαγές που σχετίζονται με την ε, απόλυση και τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, είναι ευπρόσδεκτες. Ε, τα ίδια δικαιώματα θα πρέπει να ισχύουν και για πατέρες οι οποίοι θα λάβουν, οι οποίοι θα λάβουν άδεια πατρότητας και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αρχή για να υπάρχει καταμερισμός όλων των ευθυνών ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να απολυθεί από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι και έξι μήνες ε, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας αυτή η περίοδος ε, κατά την άποψή μου θα πρέπει να αυξηθεί στον ένα χρόνο διότι οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να προσαρμοστούν και σε μια νέα εργασιακή κατάσταση και χρειάζεται κάποιος χρόνος προκειμένου να γίνει αυτό. Γι' αυτό και εγώ προτείνω ένα χρόνο. Τώρα, για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλλαγές αρκετά σημαντικές. Ε, φυσικά είναι θετικό να επιστρέψει κάποιος στην ίδια θέση εργασίας ή σε μια αντίστοιχη θέση εργασίας, αλλά πρέπει να δούμε και τι σημαίνει η ισοδύναμη θέση εργασίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι ουσιαστικά θα είναι η ίδια θέση εργασίας τόσο όσον αφορά το μισθό και όσον αφορά στα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελούνται. Η εργαζόμενοι που έχει επιστρέψει από άδεια μητρότητας ε, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ωράριο εργασίας της ή τον τρόπο εργασίας της. Η εργοδότης οι εργοδότε δεν θα πρέπει μόνο να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα αιτήματα, αλλά ε, να τα εγκρίνουν κιόλα όταν είναι αιτιολογημένα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της δική μου πρότασης και της πρότασης τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δεκτεί σχετικό αίτημα εάν είναι εύλογο και είναι σαφώς αιτιολογημένο. Τώρα, για τις υπερορίες. Προτείνω ένα νέο άρθρο, το οποίο λέει ότι οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες ε, με παιδιά κάτω των 12 μηνών, και γυναίκες ε, κατά τη διάρκεια του θυλασμού δεν θα πρέπει να εργάζονται υπερορίες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται καθόλου στο φυλασμό. Προτείνω λοιπόν ένα νέο άρθρο, το οποίο λέει ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα σε δύο ημερήσια διαλύματα για φυλασμό μέχρι το βρέφος να φτάσει στην ηλικία των 12 μηνών. Okay, thank you. Now there is Portuguese, okay. <laughs> It's... Τώρα υπάρχει πορτογαλικά. Για μένα είναι πολύ πιο εύκολο. Okay, uh, let's uh, continue. Να συνεχίσω λοιπόν. So, uh, I was talking about um, the breastfeeding Uh, Μιλούσα λοιπόν για το θυλασμό και θα συνεχίσω στα πορτογαλικά. Ε, ε, ε, eh, Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι όσον αφορά τις γυναίκες κατά την περίοδο του θύλασμου είναι πολύ σημαντικά τα όσα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ε, για τη σημασία του θυλασμού στους πρώτους μήνες της ζωής. Ε, έχουμε και το σχετικό άρθρο της Σύμβασης 183, το άρθρο 10 του, της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία λέει ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα σε ένα ή περισσότερα καθημερινά διαλύματα ή ε, αντιστοίχως μείωση του ωραρίου εργασίας για να μπορέσει να θυλάσει το παιδί της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να εγκριθεί αυτή η πρόταση τροπολογίας η οποία προβλέπει μείωση του ωραρίου εργασίας χωρίς ε, καμία οικονομική απώλεια αντιστοίχως μπορεί να είναι δύο ώρες την ημέρα ή δύο διαλύματα ημερησίως. Τώρα, όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου, η οποία είναι σημαντική σε αυτή την πρόταση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν ε, γενετικές ανομαλίες, ε, δυσπλασίες ε, και άλλα προβλήματα και οι παράγοντες αυτές, αυτοί συγγνώμη, μπορεί να πλήξουν είτε άνδρες είτε γυναίκες. Και πλήττουν πρωτίστως το έμβριο. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να προαχθεί μια προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στην πρόληψη, η οποία θα διασφαλίζει ότι θα γίνεται μία ε, κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου στον χώρο εργασίας για τους κινδύνους σε περίπτωση που προσλαμβάνονται άτομα, άνδρες ή γυναίκες, ε, σε γόνιμη ηλικία, σε ηλικία αναπαραγωγής. Αυτό δεν αναφέρεται στην οδηγία του 92 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε προβλέψει και καμία τροποποίηση στην ε, οδηγία του 92. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διευρυνθεί το όσα, να διαφερθούν τα όσα αναφορούν στην αξιολόγηση κινδύνου, η οποία θα πρέπει να γίνεται για προληπτικούς λόγους και να αφορά και στους άνδρες και στις γυναίκες δεν ε, αρκεί να γίνεται μια αξιολόγηση κινδύνου όταν ε, μια γυναίκα ε, είναι έγκυος και ο εργοδότης της λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι είναι έγκυος. διότι αυτό συνήθως γίνεται μετά από 9-10 εβδομάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ήδη αργά για να γίνει μια αξιολόγηση κινδύνου. Ένας κίνδυνο ο οποίος γνωρίζουμε δε ότι μπορεί να χτυπήσει από τις πρώτες μέρες της εγκυμοσύνης το έμβριο. Τώρα, όσον αφορά τον κοινό καταμερισμό της ευθύνης και την επέκταση της πρότασης. Μία πρόταση η οποία ε, κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να είναι μόνο ε, μία οδηγία που θα αφορά στην άδεια μητρότητας, αλλά θα πρέπει να αφορά και στην άδεια πατρότητας. Θα πρέπει να μπορούμε να συμφιλιώσουμε ε, εργασιακή και οικογενειακή ζωή, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Επίσης γνωρίζουμε ότι η κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των προτεραιοτήτων της προβλέπει ε, την προαγωγή πολιτικών οι οποίες θα έχουν ως στόχο ε, τη συμφωλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προειδοποιήσει τα κράτη-μέλη για την ε, ύπαρξη ενός ε, δημογραφικού προβλήματος. Υπήρχε και σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, δημογραφική πρόκληση και επομένως θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις διατάξεις οι οποίες ευνοούν την συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Πέραν αυτού, Αυτό που προτείνω είναι η άδεια πατρότητας, ε, ένα διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, δύο εξ αυτών υποχρεωτικές, οι οποίες δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν, θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν από τον πατέρα, από τον άνδρα, και θα πρέπει να ε, αποζημιώνονται πλήρως και όταν κατόπιν ο πατέρας θα επιστρέψει ε, στην εργασία του μετά από αυτή την άδεια θα πρέπει να χαίρει των ίδιων δικαιωμάτων ε, σε θέματα προστασίας της εργασίας του. Δηλαδή δεν μπορεί να απολυθεί κατά το διάστημα αυτό και θα πρέπει να έχει το ίδιο ευέλικτο ωράριο με την ε, γυναίκα. Και αυτό διότι ε, πρέπει μια για πάντα να ε, πάψουν να υπάρχουν στερεότυπα ε, τα οποία διαρκούν στη ζωή μας. Η γυναίκα θεωρείται εργαζόμενη υψηλού κινδύνου διότι απουσιάζει περισσότερο από το χώρο εργασίας, απουσιάζουν περισσότερο γυναίκες γιατί μένουν έγκυες και αποκτούν παιδιά. Ουσιαστικά λοιπόν θεωρούνται δεύτερης διαλογής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εμπλέξουμε και τους άνδρες στην οικογενειακή ζωή από την γέννηση του παιδιού. Θα πρέπει να ε, μοιράζονται τις οικογενειακές ευθύνες. Πέρα από την άδεια πατρότητας που είναι κάτι άλλο το οποίο θα... Ε, Ε, η οικογενειακή άδεια συγγνώμη, θα μπει σε θέματα ε, σε μια διαφορετική οδηγία. Ε, ενώ εδώ θεώρησα ότι είναι κατάλληλο να αναφέρουμε και την άδεια πατρότητας πέρα από την άδεια μητρότητας. Ζητώ συγγνώμη γιατί τα έκανα λίγο θάλασσα, είχα προετοιμάσει την ε, παρουσίασή μου στα, αγγλικά, στα πορτογαλικά, μετά υποχρεώθηκα να τα πω στα αγγλικά, κάπου χάθηκα. Ελπίζω όμως να ήμουν σαφή ω προς τις προθέσεις μου και τις προτάσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, Edit τα κατάφερες μια φορά στις δύο γλώσσες, διότι το κοινοβούλιο μας είναι γλωσσό και έτσι καταφέρνουμε να περνάμε από τη μια γλώσσα στην άλλη. Ε, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, διότι είναι θέματα που αφορούν πραγματικά και τη φύση της γυναίκας και την καθημερινή ζωή, αυτά που λέγαμε προηγουμένως ότι απασχολούν τις ε, Ευρωπαίες γυναίκες μετά τα αποτελέσματα του, της έρευνας του βαρομέτρου. Τώρα ερχόμαστε στην κυρία Στριντ Λούλινγκ, ε, η οποία θα μας μιλήσει για την έκθεση. Η οποία θα μας μιλήσει για την έκθεσή της. Je dis à Astrid que tu vas nous parler de, de ton rapport euh, sur le, euh, les pensions ou les droits à la, la sécurité sociale. Κοινωνική ασφάλεια. Συντάξεις. Θα τα πω, θα τα πω, μην ησυχείτε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι συγγήτρια για τη νέα πρόταση οδηγίας που αφορά την ισότητα μισθών ανδρών και γυναικών που ασκούν μια ανεξάρτητη δραστηριότητα. Στην αιτιολογική μου έκθεση άρχισα λέγοντας αυτή η οδηγία που έχουμε από το 86 Είναι μια οδηγία που έχει ένα μακρό, μακρύ ιστορικό, αλλά όχι και πολύ ε, καλό παρελθόν. Γιατί το κέντρο μου βιωθήκε το 86 από τους υπουργού ε, είναι χωρίς καφέινη τελείως. Και δεν φτάνει καν αυτά που είχε προτείνει η Κομισιόν το 1984. Και γι' αυτό αυτή η οδηγία δεν απέδωσε καθόλου. Γιατί σε εκθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ξεκάθαρα ότι το κείμενο αυτό δεν επέτρεψε να βελτιωθεί η κατάσταση των ανεξαρτήτων οργανωμένων και των συζύγων τους όσον αφορά την ισότητα μισθών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει εδώ και πολύ πολύ καιρό, δεν ξέρω πόσα ψηφίσματα προετοιμάσαμε στα πλαίσια των οποίων ζητήσαμε την τροποποίηση της οδηγίας αυτής. Εγώ προσωπικά το 1997 είχα προετοιμάσει μια έκθεση που ασχολούνται πλήρως της κατάστασης αυτής των συζύγων των ανεξαρτήτως εργαζομένων, γιατί τότε η κατάσταση ακόμα πιο σοβαρή από ό,τι για τους ίδιους τους ανεξάρτητους αυτοαποσχολούμενους. Γιατί αυτή η σύζυγοι, τέλο πάντων εταίροι, είναι αόρατη δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση και γι' αυτό είχαμε ζητήσει πάνω από 12 χρόνια έχουν περάσει μία τροποποίηση της οδηγίας αυτής για να μπορεί να είναι πιο περιοριστική και για να φτάσουμε σε υποχρεωτική ε, εγγραφή των συζύγων και εταίρων για να μην είναι πια όρατη και η υποχρέωση των κρατών μελών θα μέτρα ούτως ώστε οι σύζυγοι αυτοί να μπορούν να συνάψουν μία ασφάλεια για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για τη σύνταξή τους. Τέλος, η Κομισιόν έτεκε πρόταση οδηγίας που προωθεί την οδηγία του 86 και προτείνει ένα νέο κείμενο. Σας λέω όμως εκ μιας αρχής ότι δεν με αυτή η πρόταση γιατί όπως και παλιά η οδηγία έτσι και αυτή τώρα δεν θα μας επιτρέψει να λύσουμε τα πιο σημαντικά προβλήματα. Καταρχήν για να είμαι πιο σαφής θα ήθελα να μιλήσω για τους ίδιους ή τις ίδιες ανεξάρτητα εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες και μετά θα σας μιλήσω για τους συζύγους και τους εταίρους. Η ανεξάρτητη απασχόληση είναι ε, μειονοτική γιατί απασχολεί το 16% των εργαζομένων στην Ευρώπη και ένα μεγάλο ποσοστό είναι οι γυναίκες. ...71%. Έχω κι εγώ γλωσσικά προβλήματα γιατί εγώ λουξιβουργιανά είναι η μητρική μου γλώσσα. Λοιπόν, 71% των γυναικών αυτών εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών. Υπάρχουν όμως και πολλές στη γεωργία, εξίσως και άντρες, στο εμπόριο βέβαια, όλα αυτά τα, επαγγέλματα που ξέρετε ότι η που η γυναίκα είναι, κρατάται το ταμείο σε οικογενειακές επιχειρήσεις και στα ανεξάρτητα επαγγέλματα υπάρχουν πολλές γυναίκες στη γραμματεία, ας πούμε, το, μια γυναίκα που κάνει τη γραμματέα του άντρα της που είναι γιατρός και άλλων ε, ανεξαρτήτων επαγγελμάτων. Η πρώτη κομισιόν τώρα αφορά τα και τα προβλήματα δυσκολίας ένταξης, πρόσβασης των γυναικών στα επαγγέλματα αυτά και υπάρχουν προτάσεις για να διευκολυνθεί αυτή η δραστηριότητα από εκείνο το φύλλο που υποαντιπροσωπείται. Αυτό μου φαίνεται μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να προβλέψουμε και θετικές δράσεις για να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα δεξάρτητα αυτά επαγγέλματα. Μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση είναι ότι πρέπει να προβλέψουμε περιοριστικά μέτρα για να μην απαγορεύεται πια σε κανένα κράτος μέλος με το εθνικό δίκαιο η δημιουργία μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων ή μεταξύ εταίρων. Υπάρχουν ακόμη κάποιες νομοθεσίες στα 27 κράτη-μέλη όπου ένα ζευγάρι δεν μπορεί να ιδρύσει μια εταιρεία. Αυτό θα πρέπει να καταργηθεί. Και με τον, δηλαδή με τον εραστή του μπορεί κανένας να έχει μια εταιρεία, αλλά με το σύζυγο όχι. Τι είναι αυτό. Θα ήταν λοιπόν μεγάλη πλανέκτημα εδώ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε ανεξάρτητες ε, επαγγελματα. Παραδείγματος είναι κομμότριες στη γνώμη μου, στη χώρα μου. Και σε αυτή την περίπτωση, σε μια τέτοια εταιρεία μπορεί και ο και η σύζυγος να είναι μισθωτή. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ήδη αντιμετώπιση Και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να θεωρηθούν δαπάνης της εκμετάλλευσης και η μισθή των δύο. Καθώς επίσης και οι κοινωνικές εισφορές. Εκπίπνε λεπτό φορά. Αυτό είναι καταπληκτικό πρότυπο. αλλά σε ορισμένε χώρε. οι ανεξάρτητοι και οι σύζυγοι τους θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κοινωνική ασφάλεια. Δεν ξέρω, δεν μελέτησα όλους τους ογκώδεις ε, ογκώδεις μελέτες της Κομισιόν. Κατά πόσον αυτό ισχύει για τους ανεξάρτητους εργαζόμενους, ότι υπάρχει δηλαδή υποχρέωση να ενταχθούν στην κοινωνική ασφάλιση. Αν ναι, καλώς. Εάν όχι, πρέπει να το προβλέψουμε. Γιατί δεν επιτρέπεται τα άτομα αυτά να παραμείνουν χωρίς κοινωνική κάλυψη και προστασία. Και ζητήσαμε επίσης στην έκθεσή μας, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν στους συζύγους αυτούς να ενταχθούν στις τα ταμεία, δηλαδή ο, εάν υπάρχει νομοθεσία ε, εργαζόμενος να μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνική ασφάλεια, να πρέπει και ο σύζυγος ή η σύζυγος να μπορεί να ενταχθεί στο ίδιο ταμείο. Υπάρχουν ορισμένε χώρε που δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Έγινε όμως κάποιο άνοιγμα από πολλά κράτη-μέλη και πιστεύω ότι το άνοιγμα αυτό θα πρέπει να γενικευτεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή η οδηγία να προβλέπει όλοι την εξάρτητα εργοζόμενη να έχει μια κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και η σύζυγή τους να είναι επίσης στο ίδιο ταμείο. Ο χρεωτικός. Στη χώρα μου έχουμε ένα πάρα πολύ καλό, καταπληκτικό σύστημα για τους παραγωγούς, αγροτικούς παραγωγούς. Και οι δύο πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλιστούν. Όταν το 1974 πέρασε ο νόμος αυτός, ούλιαζαν. Αλλά τώρα είναι υπερευτυχής γιατί μπορούν να ωφεληθούν και οι δύο από μία σύνταξη. Για να είμαι σύντομη, γιατί πρέπει να τελειώνω από το μου λένε και έχω υποβάλει και τις σχετικέ τροπολογίες για αυτό που θέλω, δηλαδή να μην ε, είναι εθελοντική η ένταξη των συζύγων γιατί κάναμε πολλές, ε, πολλά πειράματα και στη χώρα μου υπάρχουν εκατοντάδες ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν και δεν μπορούν, δεν έχουν ενταχθεί γιατί κοστίζει. Να σας πω και δύο λόγια, με συγχωρείτε πρόεδρε, και για την προστασία της μητρότητας. Γιατί η πρόταση αυτή καλύπτει και τη μητρότητα. Η Κομισιόν προβλέπει η προστασία μητρότητας των ανεξαρτήτων απασχολουμένων να αντικατοπτρίζει την ισχύουσα οδηγία του 92 για τους μισθωτούς. Εγώ είμαι κατά. Δεν μπορεί να συγκριθούν οι ανεξάρτητοι και οι σύζυγοί τους με τους μισθωτούς. Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν είναι τελείως διαφορετικές. Και ζητάω στο κείμενό μου και είμαι κατά για αυτό της μιας τροπολογίας της κυρίας Εστρέλα που θέλει να επιβάλλει υποχρεωτική ε, διακοπή εργασίας 8 εβδομάδων σε όλους τους εργαζόμενους είτε σύζυγοι, είτε άνεργοι, είτε ε, μισθωτοί, είτε ανεξάρτητοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω προτείνει μια τροπολογία όπου δίνεται η άδεια μητρότητος σύμφωνα και με τις ανάγκες της ειδικέ των εξαρτήτων εργαζομένων και των συζύγων τους. Έχω υποβάλει και άλλες τροπολογίες, αλλά αυτό που καταμένει το πιο σημαντικό είναι αυτά που σας είπα για να αλλάξει η κατάσταση των εξαρτήτων και τα βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν γιατί πάλι η δεκαφεϊνέ ναι, είναι. Ξέρω ότι πολλές κυβερνήσεις δεν συμφωνούν. Ξέρω ότι και οι ίδιοι ανεξάρτητοι αυτοαπασχολούμενοι δεν συμφωνούν. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, ακόμα και για αυτή την πρόταση της Κομισιόν, όπου όλα γίνονται ελεύθερα, κατόπιν ετήσεως, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε ίσως να φτάσουμε σε ένα κείμενο κατάλληλο με συνένεση εδώ. Και εγώ θα ήθελα να φτάσουμε και πριν από τι εκλογέ στην υιοθέτηση αυτής της οδηγίας σε πρώτη ανάγνωση. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Αστρίτ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο για τα συμπεράσματα στην Πρόεδρο που σας είχα προαναγγείλει της Επιτροπής Γυναικών, την κυρία Ζαμπόσκα και μετά όταν θα έχετε μια πλήρη εικόνα του ρόλου της Επιτροπής Ισότητας των Ευκαιριών που ασχολείται κυρίως με τα θέματα αυτά, θα μπορείτε, λέω, να υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις. Λίγες ερωτήσεις, δεν έχουμε πολύ χρόνο στην κυρία Ζαμπόση και στις ηγητρίες. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκπρόσωποι του Eurostat, αγαπητοί συνάδελφοι. Ίσως θεωρείτε ότι είμαι πολύ παρά παράτολμη να έρθω εδώ ένα τέταρτο που κλείσει το συνέδριο για να καταλήξω σε συμπεράσματα αυτό που συζητάγατε όλο το απόγευμα. Euh, Θα ήθελα να πω δύο λόγια πάνω σε ευρωεκλογέ και την άποψη των γυναικών πάνω στο θέμα αυτό. Προσωπικά δεν ήμουν παρούσα, αλλά είχα τους συνεργάτες μου και αυτοί μου τα μεταβίβασαν τις πληροφορίες για το τι συζητήσατε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Μου είναι σημαντικό να είμαι σε διάλογο με όλους τους δημοσιογράφους που βελτιώνουν την εικόνα της ε, γυναίκας στην κοινωνία. Οι συνεργάτες μου τόνισαν κάποια σημεία όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου. βλέπω ότι ένα στους δύο θεωρούν ότι θα πρέπει το 50% των βουλευτών να είναι γυναίκες και ότι η εμπιστοσύνη είναι του Παϊκού Κοινοβουλίου και η κύρια ανησυχία των γυναικών είναι να βελτιωθεί το σύστημα της φροντίδας των παιδιών. Μπορούμε να συνεχίσουμε όλα αυτά, αλλά διαβάζοντας τα είναι πραγματικά ένας κατάλογος αποτελεσμάτων που αντικατοπτρίζει τις εργασίες της Επιτροπής των Δικαιωμάτων της Γυναικών. Πέντε σημεία έχω εδώ και ομολογώ ότι πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών έχει προετοιμάσει μία έκθεση πρωτοβουλία για αυτό το θέμα. Δηλαδή η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών με την εργασία της ε, ανεκατοπτρίζει ανησυχίες των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Γιατί προετοιμάσαμε και διάφορες εκθέσεις πάνω στις γυναίκες στον τρίτο κόσμο. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις προσωπικές. Αν θέλουμε οι γυναίκες να διαφερθούν για τις ευρωεκλογές, θα πρέπει να τους ε, ενημερώσουμε πάνω στα θεσμικά όργανα της κοινότητας και ιδίως του τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Euh, euh, Έγινε στη Σλοβακία τη χώρα μου μια δημοσκόπηση και τρέπομαι να σας το πω. Το 50% δεν ήξεραν ότι φέτος υπάρχουν ευρωεκλογέ. Και είμαι σίγουρη ότι στις άλλες χώρες, στις παλιέ χώρε τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει η εικόνα, αλλά στις νέες χώρες είναι η ίδια ε, κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να ανακοινώνουμε τις πληροφορίες στους πολίτες. Εάν θέλουμε να επικοινωνήσουμε πάνω στην πολιτική πραγματικότητα θα πρέπει να επι ε, να επιδιώξουμε να επικοινωνούμε σωστά. Δεν κάνουμε πολιτική για τους δημοσιογράφους. Δεν κάνουμε πολιτική για την καθημερινή ζωή όλων. Πρέπει να σας το πούμε. Γιατί συχνά υπάρχουν πληροφορίες σύντομες που δεν αντικατοπτρίζουν την εργασία μας. Expérience depuis le début de la législature, il faut inviter les journalistes et aussi les journalistes nationaux, non seulement les journalistes accrédités ici auprès de l'Union européenne, à, nos événements. Θα πρέπει πάντα κοινή γνώμη να είναι ενήμερη για το τι κάνουμε εδώ. Θα σας πω ότι οι δημοσιογράφοι από τη Σλοβακία που επισκέφτηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλαξαν Τελείω την άποψή του για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, ότι το θέμα της κοινωνικής ασφάλειας δεν είναι και της κοινωνικής ισότητας δεν είναι πάντα στην πρώτη σέλιδα των εφημερίδων κάθε μέρα. Δεν πρόκειται να αναζητήσω τώρα τους λόγους γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. με, οι κύριες θέσεις είναι καλύπτονται από άντρες, ίσως γι' αυτό δεν ξέρω αν αυτός ο λόγος. Όμως, η ισότητα των ευκαιριών δεν μπορεί να είναι θέμα αμφισβητήσει. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το θέμα αυτό και οι υπεύθυνοι πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες, να μην το παραβλέπουν. Γιατί καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι μιλάμε πολύ για ισότητα, χωρίς τελικά να γίνεται τίποτα. Και στην ετήσια μου εκθεσία όταν κάνω την αξιολόγηση του λεγόμενου mainstreaming φίλων ότι η ισότητα των ευκαιριών, η ισότητα ανδρών και γυναικών δεν είναι πάντα το κύριο θέμα. που τους απασχολεί. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών Θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την Επιτροπή μας. Θα πρέπει κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια και να παρουσιάζουμε την νομοθεσία μας και φέτος με τους συναδέλφους των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων η Επιτροπή ε, ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών οργανώνει αύριο μία εκδήλωση για την ημέρα των γυναικών του 2009 και σας καλώ αύριο να δείτε και να συνεχίσετε τη συζήτηση αυτή. Αύριο το πρωί στο ημικύκλιο του Κοινοβουλίου εδώ στον Τριτόροφο στις 9. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο, έχετε να κάνετε κάποια ερώτηση ουσιαστική, εύστοχη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Οι τοποθετήσεις σας μπορούν να έχουν σχέση και με τα προηγούμενα θέματα του πάνελ. Η κυρία Στρέλα είχε κάνει μια παρατήρηση. για να αιτιολογήσω την πρόταση μου τροπολογίας που ανέφερε η κυρία Λούλινγκ. Κατά τη γνώμη μου, οι υπάλληλοι ή οι άνεργες γυναίκες, ας πούμε η οδηγία για τη μητρότητα, δεν καλύπτει τις οικιακές βοηθούς. Και τη γνώμη μου, όλες οι γυναίκες χρειάζονται 6 ή 8 εβδομάδες σύμφωνα με τη γνώμη των γιατρών για να μπορέσουν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους μετά από την εγκυμοσύνη, μετά από, την, μετά από τον τοκετό. Όλες οι γυναίκες Πρέπει λοιπόν να έχουν πληρωμένες ε, ε, διακοπές από, την, ε, τον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι θέμα δικαιοσύνης, ισονομίας, απαραίτητο για να εξασφαλίσει σε όλες τις γυναίκες έναν ελάχιστο χρόνο για την ανάρρωση μετά τον τοκετό. Μόνο δύο ερωτήσεις μπορούμε Λοιπόν, ποια θέλει το λόγο, μια παρατήρηση, ένα γρήγορο συμπέρασμα, όχι. Δεν ζητώ λοιπόν για τη δεύτερη ερώτηση, ήταν σαφέστατα όλα. Αύριο το πρωί, όπως είπε η κυρία Ζαμπόρφσκα, μπορείτε να συνεχίσετε. Θα εμπλουτίσετε όλη σας τη σκέψη και τον προβληματισμό. Κύριε Λούλινγκ, μα κοιτάστε να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και γιατί δεν θέλω να ε, αντιγράψω το σύστημα των, ε, ε της ε, ε τοκετού των μισθωτών υπαλλήλων με τους ε, αυτόνομους εγώ δεν είπα ότι για τους αυτόνομους εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρχει άδεια κατόπιν αιτήματος. Στη χώρα μου οι αυτόνομοι έχουν ίδια άδεια με την με, με, με αυτή των μισθωτών, με των υπαλλήλων και η κυβέρνησή μου τα πληρώνει όλα. Ε, δεν έχω παράπονα, αλλά έχω όμως υπόψη μου ότι υπάρχουν και ε, στελέχη επιχειρήσεων, ε, γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις που δεν μπορούν να πουσιάσουν πάνω από ένα χρόνο. Ξέρετε για, τους, να, για τις μισθωτές στη χώρα μου. Αν έχετε ας πούμε την εγκυμοσύνη σας 4 ε, Μαρτίου και 12 Αυγούστου γεννάτε 12 εβδομάδες άδειας τελειώνει 8 Νοεμβρίου έρχεται επίσης και η γονική άδεια την οποία δικαιούνται και οι αυτόνομοι εργαζόμενοι 6 μήνες τέλη 2010 δηλαδή θα ξαναπάει στη δουλειά της ε, η εργαζόμενη. Εσύ πιστεύετε ότι μία επιχειρηματίας ένα χρόνο θα, θα λείπει από τη δουλειά της αν έχει ένα παιδί πρέπει να είμαστε ε, ρεαλιστές και υπάρχουν ε, και τροπολογίες της κυρίας Εστρέλα που θέλουν να εφαρμόσουν τα παραρτήματα 1 και 2 της οδηγίας που λένε ότι όταν δεν θέλετε να ασκήσετε ορισμένες εργασίες Αλλά αυτό θέλει να ισχύσει και για τους άντρες. Για τους άντρες και για τις γυναίκες ε, σε φάση αναπαραγωγής. Εμένα η μαμά μου με αναπαρήγαγε στα 42 της. Οι άντρε ακόμη παραπάνω μπορούν να αναπαραγωγούν. Είναι ανεφορίου. Λοιπόν, άμα κάνετε τέτοιες τροπολογίες και άμα κοιτάξτε και τον κατάλογο των όλων όσων θα μπορούσαν να γίνουν, τότε θα διαγράψετε πραγματικά όλους τους άντρες από τις υπόγειες εργασίες. Δεν θα, μέχρι 60 χρονών κανένας άντρας δεν μπορεί να ασκεί ε, ε, υπόγειες εργασίες διότι μέχρι τα 60 να παράγει. Λοιπόν, ας είμαστε λογικοί. Ήθελα να σας τα πω δηλαδή αυτά. Γι' αυτό εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτές τις τροπολογίες, διότι αυτές οι τροπολογίες θα στραφούν καταρχήν κατά των γυναικών των ιδίων, μετά κατά των επιχειρήσεων, διότι δεν θα είναι σε θέση να εργαστούν με αυτές τις τροπολογίες. Να, σας το λέω ειλικρινά. Τέλος πάντων θα ασχοληθούμε με το θέμα, αλλά σας το λέω εσά δημοσιογράφου και άλλε, ότι άμα υποβάλλουμε προτάσεις 12 μήνες, 24 μήνες, το ευρωπαϊκό λόμπι θέλει 24 και πάει λέγοντας. Αλλά στη χώρα μου οι γυναικείες οργανώσεις δεν θέλουν αυτή την παράταση, διότι θεωρούν ότι αυτό βλάπτει τις ίδιες τις γυναίκες. Διότι οι εργοδότες διστάζουν όλο ένα και περισσότερο να απασχολούν οι γυναίκες. Θα σταματήσω εδώ διότι ήθελα απλώς να σας περάσω αυτό το μήνυμα. Διότι όλοι βρισκόμαστε ε, εδώ υπό την ίδια σκέπη και ψάχνουμε να δούμε τι είναι πιο ρεαλιστικό και για τις γυναίκες και για την οικονομία. Ευχαριστώ Άστριντ, ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας. Πραγματικά μας ενθαρρύνετε. Διότι είμαστε πεπισμένες ότι θα έχουμε τη συνεργασία σας και μετά τις 8 Μαρτίου και κατά την προκλογική εκστρατεία που θα μας βοηθήσετε να προβάλλουμε το ρόλο της γυναίκας, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ρόλο της γυναίκας μέσα στο Κοινοβούλιο και τις εμπνεύσεις τους. Λοιπόν, θα πιούμε τώρα ένα ποτήρι στην υγεία και στο κουράγιο των γυναικών.